Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε εκ νέου τη συνεδρίασή μας. Σήμερα το απόγευμα έχουμε τους δύο Πολωνούς ε, υπουργούς, ε, τον Υπουργό Μεταφορών και στη συνέχεια τον Υπουργό Τουρισμού. Καταρχάς λοιπόν με τα χαράς καλωσορίζουμε τον ε, Υπουργό Γκραμπάτσης Ελπίζω να πέτυχα λίγο την προφορά του ονόματά σας, έστω και λίγο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας για την ε, Επιτροπή Μεταφορών και κατόπιν ο συνάδελφός σας, η συνάδελφός σας, συγγνώμη, η κυρία Σαμπριάσκα, θα κάνει την παρουσίαση του τουρισμού. Καταρχάς λοιπόν σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Υπουργέ. Προσβλέπουμε με ανυπομονησία στα όσα θα μας πείτε και έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Την 1η Ιουλίου η Πολωνία με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβε τα ενία την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η χαρά συνοδεύεται από ιδιαίτερη, ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη συνέστηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεδομένης αυτής της δύσκολης κρίσης που βιώνουμε. Εμείς την Προεδρία αυτή την προετοιμάσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα και υπήρξαν και πολλές ε, συναντήσεις. Ε, έχουμε πέρα από αυτό και συναντήσει και είχαμε επαφές και με τους συντονιστές και τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Συναντηθήκαμε με πολλούς και πολλές ε, ώστε να προετοιμάσουμε την Προεδρία μας. Την πρώτη συνάντηση της Προεδρίας μας την είχαμε ήδη κατά την διεξαγωγή της προηγούμενης Ολομέλειας στην περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαμε σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν που κατέστησαν εφικτό το να μπορέσουμε για παράδειγμα να αντιμετωπίσουμε το θέμα των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των ποινών που πρέπει να επιβάλλονται. Και τώρα θέλουμε να παρουσιάσουμε τα μέτρα, της προτάσεις ε, το σχέδιο, το πρόγραμμα της, Ευρωπαϊκής, της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Κανείς δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι τα θέματα μεταφορών έχουν μεγάλη προτεραιότητα. Χωρίς αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών ούτε η ευρωπαϊκή οικονομία ούτε οι οικονομίες των κρατών μελών μπορούν να αναπτυχθούν και ούτε θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα με τους ανταγωνιστές τους. Ακόμα και οι πολίτες ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν τα ευρωπαϊκά αυτά διευρωπαϊκά δίκτυα για να μπορούν να μετακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια. Όταν εργαζόμαστε για την κατάρτιση του προγράμματος της Πολωνικής Προεδρίας προσπαθούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Πολωνική Προεδρία θέλει να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αναμένουμε ένα έγγραφο το οποίο θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτά τα δίκτυα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα έχουμε ένα τρίμηνο ως περίοδο ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο με τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε την αυτή Προεδρία ότι δεν είναι μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Και σε σχέση με την ε, δημοσίευση αυτών των εγγράφων έχει προηγηθεί σημαντικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε βάθος συζητήσει ε, με τα κράτη-μέλη. Η Πολωνική Προεδρία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε η επικαιροποίηση αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων να διασφαλίσει τις ε, υποδομές, να υπάρχει ένα συναφές ολοκληρωμένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν οι κυριότεροι άξονες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή συγκυρία η Ευρώπη να μπορέσει να εξέλθει, να διεξέλθει από αυτή την κρίση γοργά. Ιδιαίτερα θέλουμε την προσπελασιμότητα αυτών των ε, διευρωπαϊκών δικτύων να την βελτιώσουμε σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε οι τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν, κυρίως στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Και πέρα από αυτό θέλουμε τα ουσιώδη, τα ουσιοδέστερα δίκτυα και τα παραπληρωματικά συμπληρωματικά δίκτυα αλλά και οι διεθνείς διασυνδέσεις να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα ως προτεραιότητες και μέσα από την παρουσίαση και έγκριση του, των γενικών θέσεων μπορούμε να προχωρήσουμε. Τα θέματα που συναρτώνται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι οι διασυνδέσεις με τρίτες χώρες η Πολωνική Προεδρία θέλει έντονα και εντατικά να εργαστεί σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονικών ομόρων κρατών. Στόχος μας είναι τα συμπεράσματα του της Προεδρίας από πλευράς της Πολωνικής Προεδρίας τον Οκτώβριο να μπορέσουν να προωθηθούν και να εγκριθούν. Στις ναυτιλιακές μεταφορές η Πολωνική Προεδρία επιθυμεί το έργο στο πακέτο για την κοινωνική ημερήσια διάταξη, τα κοινωνικά θέματα στο θεματολόγιο της ημερήσιας διάταξης να προαχθούν, να μπορέσουν να διαβιβα... μόλις μπορέσουν να διαβιβαστούν αυτά τα έγγραφα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε το δυνατόν γοργότερα να επιτευχθεί πρόοδος επ' αυτών των μέτρων. Για το πακέτο των κοινωνικών μέτρων και τα ναυτιλιακά ανήκουν τα εξή στοιχεία. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κοινωνικά θέματα στην ναυτιλία, πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας των ελάχιστων προδιαγραφών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών, η αντίστοιχη δηλαδή οδηγία για την εκπαίδευση κατάρτιση ναυτικών και η εφαρμογή και οι προϋποθέσεις που θα απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του ναυτικού, σύμβαση άσκησης του επαγγέλματος ναυτικών. Ένα σημαντικό στοιχείο της Πολωνικής Προεδρίας μέσα σε αυτό το συνολικό πακέτο είναι η επανεπεξεργασία της ε, οδηγίας ε, για τις ελάχιστες απαιτήσει για την κατάρτιση και εκπαίδευση των ναυτικών βασιζόμενη πάντα στην σύμβαση του IMO. Ε, Είχαμε υπόψη τον Ιούλιο να υποβληθεί αυτό το έγγραφο. Τώρα γνωρίζουμε, μας ανακοίνωσαν ότι θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει με βάση αυτά τα στοιχεία να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση. Σημαντικό είναι για την κατάρτιση των ναυτικών να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην άσκηση του επαγγελματός τους. Στόχος της Πολωνικής Προεδρίας είναι κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου εφέτος να εγκριθεί μια γενική τοποθέτηση επ' αυτού του θέματος ως συμπέρασμα. Θέλουμε ως Πολωνική Προεδρία το έργο των προηγουμένων Προεδριών, ιδιαίτερα της Βελγικής Προεδρίας και της Ουγγρικής Προεδρίας, να το συνεχίσουμε σε σχέση με την τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλεια στις ναυτικές μεταφορές. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια αποσαφήνιση και διεύρυνση του φάσματος αρμοδιοτήτων αυτής της ε, υπηρεσίας, αυτής της οργάνωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η μέχρι σήμερα εργασία τον Ιούνιο του 2011 εγκρίθηκε με συμπεράσματα από πλευράς του Συμβουλίου με μια γενική προσέγγιση για αυτό το έγγραφο. Το, η εργασία έχει ξεκινήσει και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. αρχές Ιουνίου είχαμε το πρώτο σχέδιο του εισηγητού που υπευλήθη. Το Συμβούλιο έχει καταθέσει, έχει κάνει κάποιε τροποποιήσει σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Στόχο ήταν καταρχήν αποσαφήνιση των όρων και τη κατεύθυνση και αποσαφήνιση του πνεύματο αυτού του εγγράφου. Πρέπει να δούμε εδώ τι θεμελιώδει και τι δευτερογενεί υποχρεώσει σε σχέση με, αυτό το, με αυτή την εργασία. Για το Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει πρόσθετη αξία όσον αφορά το έργο, την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και σε σχέση με την, ε, το έργο των άλλων οργανισμών αποφεύγονται επικαλύψεις και από πλευράς ε, του εγγράφου ε, δόθηκε ιδιαίτερη ε, σημασία σε αυτή την αποσαφήνιση. Είναι ένα καλό σημείο για την εκκίνηση, για την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Πολωνική Προεδρία θέλει πέρα από όλα αυτά να συνεχίσει αυτό το θέμα έντονα και εντατικά να ε, συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει φυσικά από κοινού να αποφασίσουμε και να δούμε αν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Σε επίπεδο του Συμβουλίου επιθυμούμε ή ελπίζουμε να υπάρξει πολιτική συμφωνία το Δεκέμβριο. Και τώρα στρέφομαι στι εναέριε μεταφορέ. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε μια προτεραιότητα ως Πολωνική Προεδρία. Η προτεραιότητα αυτή είναι το πακέτο για τους αερολιμένες, για τα αεροδρόμια πάντα ευθυγραμμιζόμενοι με την ανακοίνωση, με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχουν προταθεί, τον Οκτώβριο περίπου θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πακέτου μέτρων για τα αεροδρόμια που θα βασίζεται στα εξή νομοθετικά στοιχεία. Πρώτον, ένας επιμερισμός, ένας καταμερισμός των slots για τα διαφορετικά αεροδρόμια, υπηρεσίες εδάφους, καθώς επίσης καταπολέμηση ηχητική όχλησης, καθώς επίσης και ανακοίνωση για το δυναμικό των αεροδρομίων. Η Προεδρία κυρίως θα εστιαστεί σε μια ανανέωση των προδιαγραφών και διατάξεων για τις επιδάφιες ε, ε, υπηρεσίες, υπηρεσίες ε, εδάφους θέλουμε ως Προεδρία να, σημειωθεί, να μια έκθεση προόδου επ' αυτών στις 12 Δεκεμβρίου να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο και να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα συμπεριλαμβάνει του, τον ενιαίο ευρωπαϊκό εθέρα, Single European Sky μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ενιαίων ευρωπαϊκών ουρανών έχουμε και την εντολή, το σχέδιο εντολής για την ε, ε, διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Eurocontrol. Αυτή η εντολή μπορεί στη συνέχεια σε σχέση με τη συνάντηση του ε, Συμβουλίου ελπίζουμε στις 12 Οκτωβρίου να εγκριθεί και να προχωρήσουμε. Τον Οκτώβριο επίσης αναμένουμε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κοινού με τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση και την διαχείριση της ε, έναρξης της τρίτης φάσης του εγχειρήματος ΣΕΣΑΡ. Single European Sky ε, και αυτή την χρονική στιγμή η Προεδρία θέλει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να μπορέσουν να υποβληθούν που ελπίζουμε θα εγκριθούν το Δεκέμβριο. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη διαπραγμάτευση αυτή της συμφωνίας με τρίτα κράτη θα την υποστηρίξουμε, ιδιαίτερα με ε, χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Ε, έχουμε ιδιαίτερα εδώ υπόψη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναλάβει εντολή ώστε για τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα και Αζερβαϊτζάν να προχωρήσει. Και η Πολωνική Προεδρία ενδιαφέρεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για, τις, ε, για τα θέματα για την συμφωνία, για τις εναέριες μεταφορές, ε, θέμα, θέματος επί του οποίου ε, πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εντολή που έχει με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Για τις χερσές μεταφορές. Η Πολωνική Προεδρία θέλει το σημαντικό θέμα της αναθεώρησης του πακέτου μέτρων για τους σιδηροδρόμους να το προαγάγει Ξέρετε ότι τον Ιούνιο το Συμβούλιο υιοθέτησε μια γενική θέση, τοποθέτηση για αυτό το θέμα, ήταν αρκετά δυσχερέ το εγχείρημα. Θεωρεί η Πολωνική Προεδρία ότι είναι θετική αυτή η αφετηρία για να καταλήξουμε σε μια πιο διαφανή ρύθμιση των σιδηροδρόμων και να καταλήξουμε σε μια τόνωση, μια ενδυνάμωση των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με άλλους φορείς. Στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία ε, στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο και είμαστε ταυτόχρονα πρόθυμοι για συζητήσεις και διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε στενή συνεργασία με αυτό να μπορέσουμε να προβούμε στην έγκριση αυτού του εγγράφου ήδη κατά τη διάρκεια των προκατακτικών εργασιών για την Προεδρία μας ασχοληθήκαμε ήδη με, είχαμε επαφή ήδη με την εισηγήτρια και είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση σε επικοδομητικό πνεύμα. Γι' αυτό ευελπιστώ ότι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να στεφθεί με επιτυχία και σε σχέση με το θέμα των Άλπαιων και το πακέτο για τις Άλπεις. Η Πολωνική Προεδρία εργάζεται περαιτέρω για την ε, τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά τους ταχογράφους ε, οχημάτων, φορτηγών ε, οχημάτων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί με στόχο η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών ταχογράφων, ταχογράφων να βελτιωθεί και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι ο χρόνος εργασίας επαγγελματιών οδηγών και ο χρόνος ανάπαυλας ή ανάπαυσης θα μπορεί να τηρείται και να είναι σεβαστός. Είναι ένα σημαντικό έγγραφο διότι καθορίζει τους όρους εργασίας, τους όρους απασχόλησης για τους επαγγελματίες οδηγούς και ε, θέτει το πλαίσιο για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές. Ε, στόχος της Προεδρίας είναι να ξεκινήσουν οι εργασίε στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου και φυσικά αυτό εξαρτάται επίσης από το ποιοι ρυθμοί θα ακολουθηθούν, πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε. Επιθυμούμε όμως για την σύνοδο του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου να υπάρξει μια γενική τοποθέτηση από πλευράς μας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά τις αρχές Σεπτεμβρίου η Πολωνική Προεδρία μια άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών ε, Μεταφορών ε, προβλέπει να διοργανώσει όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο θέμα αυτής της ε, συνόδου θα είναι τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα κονδύλια εκτός ε, προϋπολογισμού, πώς μπορούν να κινητοποιηθούν και είμαι πεισμένος ακράδαντα ότι στη σημερινή συγκυρία κρίσης που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοια συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα έχει σίγουρα την αξία του για τις έξω ε, προϋπολογιστικές δυνατότητες από πλευράς δομών και κονδυλίων είναι ιδιαίτερη σπουδαιότητα θέμα και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θετική ανταλλαγή απόψεων και αυτό θα καταστήσει εφικτό σε αυτό το θέμα να εξευρεθούν καινοτόμε λύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις. Κυρίε και κύριοι, εδώ και 7 χρόνια είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Πολωνία. Την Προεδρία στο Συμβούλιο την αναλαμβάνουμε για πρώτη φορά παρθένο έδαφος για μας. Πραγματικά με έντονο και εντατικό πνεύμα ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία μας για αυτή την Προεδρία. Πιστεύουμε στην καλή θετική συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και πιστεύουμε επίσης ακράδαντα ότι από κοινού μπορούμε να επιλύσουμε πολλά προβλήματα. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Minister, thank you very much for your... Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίασή σας και θα ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τον κύριο Γκρός από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μόλις μας δώσατε και σας εύχομαι και εγώ επίσης ε, κάθε επιτυχία, πολλή επιτυχία διότι αυτά που έχετε αναλάβει είναι πραγματικά ένα γενναίο, θαραλέο πρόγραμμα και γνωρίζετε επίσης ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι σύμμαχό σα, βρίσκεται στο πλευρό σας. Σήμερα ίσως ακόμα πιο πολύ από ό,τι στο παρελθόν. Διότι πραγματικά επιθυμούμε ως Ευρωκοινοβούλιο το Συμβούλιο συνολικά με τη δική σας βοήθεια να αναπτύξει ευρωπαϊκά αντανακλαστικά για αυτά τα οποία βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Και εδώ φυσικά η οικονομία διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σημαντικά χαρτοφυλάκια σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε. Και φυσικά εδώ έχουμε και μια ιστορία που πριν από το δικό σας κράτος μέλος ε, έχει απασχολήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα πέμπτης το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε μειωμένο αριθμό προγραμμάτων αλλά με αποτελεσματικό τρόπο να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, δραστηριοποίησης. Έργο μας θα είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνουμε αξιόπιστοι σε αυτή τη συζήτηση και ο ρόλος σας θα είναι πολύ σημαντικός. Αξιόπιστοι θα είμαστε όταν δεν θα χρειάζεται να συζητήσουμε 20 χρόνια για μια προτεραιότητα που πρέπει να υλοποιηθεί και δεν υλοποιείται, είτε λόγω έλλειψης βούλησης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτές οι πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λοιπόν, για να παραμείνουμε αξιόπιστοι, θα πρέπει να είναι κέντρο βάρους ε, στο Λευκό Βιβλίο, όπως και εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να προχωρήσουμε και Θέλουμε να αναζητήσουμε τη συνεργασία μαζί σας, γιατί θέλουμε πολύ χειρόπιαστα, εξειδικευμένα για τα επόμενα δέκα χρόνια να δραστηριοποιηθούμε και να θέσουμε κέντρα βάρους και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστείτε και εσείς Σε εναερίε μεταφορές. Φυσικά έχουμε τα αεροδρόμια, τους αερολιμένες και το πακέτο που θα αντιμετωπίσουμε και με τις υπηρεσίες εδάφους δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για σας. Ελπίζουμε ότι αυτά τα οποία θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία επιτυχία. Να έχουμε καλύτερη, αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών και να μην αφήσουμε την αγορά να ρυθμίσει τα πάντα. Για τις ενεργείς μεταφορές θέλω σύντομα να αναφερθώ σε κάποια θέματα. Πρώτον, αυτά τα μπλοκ της κατηγορίας των FAPS είναι σημαντικό για μας τα τα μέτρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο να σημειώσουν πρόοδο. Και αυτά τα οποία αναφέρθηκαν πιο πριν και είπα για την Ουγγρική Προεδρία, θα ήθελα να παρακαλέσω ίσως και η Πολωνική Προεδρία να θέσει ένα μήνυμα, να στείλει ένα μήνυμα, να σηματοδοτήσει ότι κατά την δική σας περίοδο, κατά τη δική σας προεδρία να μπορέσει να προαχθεί το θέμα της υπογραφής και έγκρισης αυτού του εγχειρήματο. Θα ήταν πολύ θετικό αυτό το μήνυμα, διότι θέλουμε το χρονοδιάγραμμα που έχετε ενώπιόν σας να τηρηθεί. Ένα δεύτερο θέμα για αυτή τη συζήτηση που είχαμε δύο φορές σήμερα σε σχέση με την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Εμείς αναμένουμε από το Συμβούλιο μια σαφή τοποθέτηση και δεν θέλουμε για άλλη μια φορά να ξαναζήσουμε αυτό το οποίο ζήσαμε φέτος, ότι για τελευταία στο τελευταίο λεπτό θα πούν κάποια κράτη, για παράδειγμα, ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν κάποιες προτάσεις και να πορευθούν από κοινού μετά. Αλλά είμαστε πρόθυμοι να προβούμε σε αυτή τη συζήτηση μαζί σας και είναι μια ερώτηση που προαναγγέλλω και για το τέλος της δικής σας Προεδρίας. Θέλουμε πριν από τα τέλη του 2011 μέχρι την έναρξη του 2012 να ξέρουμε τι θα γίνει. Θα είναι οι χώρες σε θέση μέχρι το 2013 που εκπνέει προθεσμία καταληκτικά να επιτελέσουν αυτό το έργο. Στις μεταφορές έχετε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρτοφυλάκι όσον αφορά τα θέματα των ταχογράφων. Οι δικέ μας απόψει για αυτόν τον τομέα είναι ότι οι ταχογράφοι φυσικά συνεισφέρουν στην ασφάλεια, για την ασφάλεια. Φυσικά καθορίζουν και βελτιώνουν τους όρους εργασίας των ε, ο επαγγελματιών οδηγών. Πρέπει όμω να είμαστε και ρεαλιστικοί και να λάβουμε υπόψη ότι διασυνοριακά <clears throat> για κάποιες ε, περιοχές και περιφέρειες έχουμε κάποιες που είναι πολύ αυστηρές, άλλες που είναι λιγότερο αυστηρές, περισσότερο χαλαρές. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνάφεια. Να είμαστε όλοι με το ίδιο πνεύμα να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Καλό θα ήταν αυτό και σε σχέση με τρίτες χώρες, σε σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διαμορφώσουμε αυτές τις σχέσεις με θετικό, σε θετικό πλαίσιο. Τα βιώματά σας είναι θετικά, η δική σας εμπειρία. Χαιρόμαστε λοιπόν για την δική σας προεδρία και προσβλέπουμε Βλέπουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ελκαντράου από τους Σοσιαλιστές έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς εκ μέρου τη ομάδας μου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Μας απαριθμίσατε ένα μακρύ κατάλογο θεμάτων Βέβαια για πολλά από αυτά ε, πρώτα απ' όλα πρέπει κάτι να προτείνει η Κομισιόν. Είναι ίσως ηρεμία πριν την καταιγίδα, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αυτό είναι σαφές. Δεν θέλω να καλύψω τα πάντα, θα επιμείνω σε δύο-τρία θέματα που θεωρώ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ενέργειες μεταφορές, που αποτελεί προτεραιότητα, όπως είπατε, της Προεδρίας σας Φυσιολογικό αυτό από τη στιγμή που έχουμε τη δέσμη των μέτρων των αερολιμενικών. Είπατε επίσης για το Σέζαρ και σε ό,τι αφορά το Single Sky, τον ενίο, ουρανό, θέλω να σας πω ότι όπως και ο προλαλής σας συνάδελφος και εγώ ανησυχώ για το κατά πόσον μέχρι το τέλη του έτους 2012 ε, θα μπορούν τα κράτη-μέλη να καταστήσουν επιχειρησιακά λειτουργικά αυτά τα FABs, τα Functional Airspace Blocks. Και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε αυτό το θέμα γιατί αυτό είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνιστά οικονομίες κλίμακας και βοηθά επίσης και σε ό,τι αφορά την ε, ρήπανση. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα πάνω σε αυτό το θέμα και να εκπέμψετε σαφή μηνύματα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι της, ε, των αεροπορικών μεταφορών, η ασφάλεια, μιλήσατε για αυτήν, αλλά δεν μιλήσατε για τις οδηγίες ε, που ε, άπτονται των θεμάτων χρηματοδότησης της ασφάλειας. Αυτό το θέμα το διαχειρίζεται ο συνάδελφος Γιώργ Λάιχτφριντ, ο συνάδελφός μας, και έχει παγώσει στο Συμβούλιο εδώ και κάποιο καιρό, είναι στο ψυγείο. Θα το βγάλετε εσείς από το ψυγείο, έχετε αυτή την πρόθεση. Τώρα, θαλάσσιες μεταφορές. Νομίζω ότι πράγματι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις για την ε, κοινωνική θαλάσσια ατζέντα. Είναι και προτεραιότητα για τη δική μας ομάδα. Ο συνάδελφος ε, Φλέκενστάιν φαντάζομαι θα πει τα σχετικά στο πλαίσιο και της δικής του έκθεσης. Μιλώ για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας και για άλλα θέματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των μεταφορών, τα TEN-Ts, εισερχόμαστε σε μια πολύ σημαντική περίοδο γιατί πρέπει να σχεδιάσουμε το γεωγραφικό χάρτη με τους διαδρόμους, τους άξονες, τα αεροδρόμια, τους λιμένες κτλ. Αυτός θα είναι ο πυρήνας ε, του δικτύου, αλλά πρέπει να είμαστε και συνεπείς. Τι εννοώ. Δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε όλα αυτά να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει να βρεθεί χρηματοδότηση. Να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Και βέβαια ξέρουμε ότι όλα αυτά συμπίπτουν χρονικά και με τη συζήτηση για το προπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και όπως καταλαβαίνετε, σε ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές, εμείς θα τονίσουμε ε, τα προγράμματα εκείνα, τα έργα εκείνα τα οποία συνιστούν για μας υπεραξία. Έχουν μια προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Είμαστε επίσης υπέμαρχοι της αρχής use it or lose it, όπως ε, λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, δίνουμε πόρους για την υλοποίηση ενό προγράμματο, ενό έργου, αλλά χάνονται για το κράτο μέλο ε, τα κονδύλια αυτά αν δεν έχει υλοποιηθεί εντό των προθεσμιών. Και μπαίνουν στο Ταμείο Μεταφορών τα κονδύλια αυτά, τα οποία αλλιώ θα τα χάναμε. Και ένα τελευταίο θέλω να αναφέρω για τον προπολογισμό. Δεν είναι δική σα άμεση αρμοδιότητα, το γνωρίζω αυτό, αλλά θέλω να σα ε, ζητήσω με του συναδέλφου σα από τον προπολογισμό, από τον τομέα τη οικονομία, να σκεφτείτε λίγο και να προασπίσετε όλα όσα έχουν να κάνουν στις μεταφορές. Διότι τώρα πράγματι έχουμε την πρόταση της Κορεπέρ για τον προπολογισμό του 2012. Σε αυτή την πρόταση για τα διευρωπαϊκά των μεταφορών προβλέπονται εξοικονομήσεις 101 εκατομμύριων ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία πλευρά να θέλουμε φιλόδοξο δίκτυο και από την άλλη πλευρά ε, να εξοικονομούμε ή να θέλουμε να εξοικονομήσουμε 101 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σας το λέω εν παρόδο, αλλά σας ζητώ να προσέξετε πάρα πολύ το θέμα αυτό και το ίδιο ακριβώς ε, ισχύει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα διατύπωσε τι προτάσει τη και έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση την οποία θα κάνουμε για αρκετά χρόνια πιστεύω. Ελπίζω και εσεί να φροντίσετε τα συμπληρωματικά κονδύλια που προβλέπονται από την Κομισιόν για τι μεταφορέ να μείνουν στον προπολογισμό. Ελπίζω να προβλέπετε να υπάρχουν αρκετέ ευρωπαϊκέ πιστώσει ώστε να επενδύσουμε στι μεταφορέ μέχρι το 2020. Θα μείνω εδώ. Εθίγησαν και κάποια άλλα θέματα. Νομίζω τα σημαντικότερα τα ανέφερα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Κυρία Μπιλμπάου τώρα από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να απαντάμε σε όλες τις προσκλήσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για όλα όσα μας είπε. Να πω καταρχάς ότι συμφωνούμε και είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε την οδηγία για την κατάρτιση των ναυτικών. Ε, είναι και πολύ επίκαιρη διότι ε, γίνεται και αναθεώρηση της ΕΜΣΑ. Στην ΕΜΣΑ υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που αναφέρονται και στην ε, κατάρτιση των, ε, των ναυτικών για να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα. Συμφωνούμε λοιπόν με την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, διότι θεωρούμε ότι θα βελτιώσει όχι μόνο την κατάσταση των ανθρώπων που εργάζονται στη θάλασσα, αλλά έχει και στενή σχέση με την ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα το πακέτο των αεροδρομίων, η πολιτική μας ομάδα ανυπομονεί να αναλύσει το περιεχόμενό του, αλλά θεωρούμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες για τη δέσμη των μέτρων για τα αεροδρόμια θα πρέπει να ε, συνάδουν και με όσα εκκρεμούν. Ε, το λέμε συνεχώ και λέμε ότι θα πρέπει να δώσουμε και μια τελευταία όθηση για να δημιουργήσουμε αυτό τον ενιαίο ουρανό επιτέλους και να βρούμε κατάλληλες αποτελεσματικές λύσεις για περιπτώσεις και καταστάσεις οι οποίες είναι προβληματικές. Χαιρετίζω και συμφωνώ μαζί σας ως προς το γεγονός ε, ότι οι συμφωνίες με τρίτες χώρες τις οποίες ε, αναφέρατε το Αζερβαϊτζάν, ε, η Ουκρανία και η Βουλγαρία είναι πολύ ενδιαφέρουσες για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε τέτοιες συμφωνίες. Τώρα, η πρώτη δέσμη ε, σιδηροδρομικών μέτρων. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε λύση. Είδαμε και τι γίνεται με τη συζήτηση που έχουμε αυτές τις μέρες για τη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Ε, σας ε, προτρέπω λοιπόν να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι για να διασκεδάσετε αμφιβολίες και να προσεγγίσετε θέσεις και θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι ημερομηνίε κλειδί για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτή την πρώτη δέσμη μέτρων για τα σιδηροδρόμους. Θα ήθελα να μας πείτε μέχρι πού θα θέλατε να φτάσουμε, ώστε να δούμε και τι θέση μπορούν να λάβουν οι διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες ε, εδώ. Θα έχουμε τώρα και μία αναθεώρηση με ε, περικοπές στον προπολογισμό και θέλουμε να σκεφτείτε ε, καινοτόμα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων αυτών. Οι φιλελεύθεροι έκαναν και κάποια εργαστήρια, κάποια σεμινάρια όπου είδαμε ότι η σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ε, καινοτομίες που θα συνεχίσουν να μας βοηθούν να ετοιμάζουμε υποδομές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ε, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για τον τουρισμό να σας πω ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε κι εσείς να δώσουμε μια όθηση και να δώσετε κι εσείς μια όθηση από πλευράς Προεδρίας διότι ο τουρισμός είναι προτεραιότητα της πολιτικής μας ομάδας των φιλελευθέρων και διότι η Ευρώπη έχει μεγάλες δυνατότητες οι οποίες θα επιτρέψουν μέσω του τουρισμού να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας, εάν γίνει με το σωστό τρόπο. Εν κατακλείδη, όσον αφορά την αγορά των σιδηροδρόμων, δεν αναφερθήκατε στις ε, σιδηροδρομικές εταιρείες και δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει επί τούτου ή είναι κάτι ε, το οποίο δεν θα σας απασχολήσει ε, στο μέλλον ε, και αυτό θα ήθελα να το συσχετίσετε και με τη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπάου, να σας υπενθυμίσω ότι ο Υπουργό Τουρισμού θα έρθει αργότερα. Επομένως, τα θέματα του τουρισμού μπορείτε να τα απευθύνετε στην Υπουργό Τουρισμού. Να ζητά συγγνώμη κυρία Παραντίκα. Ο κύριος Βαντάλερ από την Ευρώπη των Συντηρητικών και Δημοκρατών. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Σας ε, καλοχαιρετίζουμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια προς την Πολωνική Προεδρία. Πολύ πρωτότυπο ότι ξεκινήσατε με τη διανομή φραουλών. Σύμφωνα με την αρχή, τα πολωνικά έχουν την καλύτερη γεύση, τα πολωνικά προϊόντα και λόγω ε, κάποιας αλλεργίας δεν μπόρεσα να απολαύσω. Ήταν όμως μια εξαιρετική θα έλεγα αφετηρία, με εξαιρετική κίνηση ως πρωτοβουλία και καλή συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να αναφέρω το πρώτο το οποίο με ενδιαφέρει, ναυτιλιακές μεταφορές Είναι καλό το ότι το έχετε θέσει πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει πάντα να σταθμίζουμε τα θέματα ασφάλειας και απασχόλησης βέβαια. Εν πάση περιπτώσει και μια άλλη πτυχή προστίθεται σε αυτά τα θέματα και θέλω να την αναφέρω αυτήν εδώ. Και αυτή αφορά φυσικά το θελκτικό, ελκυστικό χαρακτήρα αυτού του επαγγέλματος. Πολλοί ναυτικοί προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρώπης και αυτό έχει επιπτώσεις στην βιομηχανία αυτή, ας την αποκαλέσουμε έτσι. Και τα όσα συμβαίνουν στις ε, δραστηριότητες ε, της, ε, του θαλασσινού, του ναυτικού επαγγέλματος πρέπει να μας απασχολήσουν. Και φυσικά η όρια απασχόλησης και η θελκτικότητα, ο χαρακτήρας είναι σημαντικά στοιχεία για αυτό το επάγγελμα. Μέσα στο πλαίσιο του πακέτου αυτού δεν αναφέρατε τα πάντα φυσικά, δεν ήταν εξαντλητική η ε, αναφορά. Τώρα για τις ναϊάδες. Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται καθοδόν αυτό το πακέτο μέτρων. Θα μπορούσατε όμως να ενθαρρύνετε για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αυτό το πακέτο μέτρων έγκαιρα να προταθεί και να υποβληθεί όσον αφορά τις ε, ποτάμιες πλωτές μεταφορές. Ε, θα ήθελα κάτι να ακούσω για αυτό το θέμα. Ήδη έχετε ίσως ε, ενημερώσει και πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στη συνέχεια διευρωπαϊκά δίκτυα. Εξαιρετικό να μιλάμε για αυτά, να ανταλλάσσουμε απόψεις, αλλά όλοι γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή την περίοδο περνάμε μια τεράστια κρίση που βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν καθημερινά οι Υπουργοί Οικονομικών ε, συνέρχονται και διαβουλεύονται πώς μπορούμε να διεξέλθουμε από αυτή την κρίση. Τι θα γίνει και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει μια θετική συνέχεια με βάση τα όσα εσείς αναφέρατε για να μπορέσει να υπάρξει ένας πυρήνας ε, δικτύων από τα συνολικά αυτά σχέδια να δούμε τι θα ενταχθεί σε αυτόν τον πυρήνα και τι δεν θα ενταχθεί. Παρακαλώ λοιπόν να παραμείνουμε πιστοί σε αυτές ε, τις αρχές ε, για αυτόν τον πυρήνα έργων και να μην εξαιρεθούν ή αφαιρεθούν πολλά. Να παραμείνουμε σε έναν πυρήνα που να αξίζει τον όρο πυρήνα ώστε να έχουμε από την άλλη πλευρά θάρρος να πούμε όχι σε τεράστιους καταλόγους ευχολόγια επιθυμιών, κρατών μελών αλλά να προχωρήσουμε με ένα πυρήνα αποτελεσματικό εναέριες μεταφορές. Τώρα το πράσινο βιβλίο για το μέλλον των εναέριων μεταφορών, καθώς επίσης και από την άλλη πλευρά και η Επιτροπή Μεταφορών ακολουθούν μια μεγάλη κατευθυντήρια γραμμή, δηλαδή μια κατεύθυνση πώς μπορούμε να πρασινίσουμε περισσότερο τις μεταφορές, να, κάνουμε, ε, να έχουμε μεταφορές που θα είναι πιο καθαρές για το περιβάλλον, θα επιβαρύνουν λιγότερο ηχητικά το περιβάλλον, αλλά και λιγότερο με ρήπους, ε, με τις εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, για να μπορέσουμε τις πιο καθαρές και πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές να προαγάγουμε. Είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για την προαγωγή αυτών των μεταφορών. Πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα. Να δημιουργηθούν λοιπόν κίνητρα ώστε να καταφέρουμε να επενδύσουμε, να υπάρξουν επενδύσεις που θα διασφαλιστούν για οχήματα, είτε είναι αυτά αεροπλάνα είτε άλλα, που θα εκπέμπουν, θα εκλείουν στην ατμόσφαιρα λιγότερους ρήπους και χερσαίες μεταφορές στο τέλος τέλος. Τίθεται το ερώτημα για μένα. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες προδιαγραφές και ρυθμίσεις ε, και διατάξεις. Σημαντικότερο θα ήταν, πιστεύω εγώ, να διαρωτηθούμε πώς οι υφιστάμενες ή ενισχύ σήμερα διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Έχουμε διαφορές σε σχέση με την εφαρμογή, την υλοποίηση. Εκείνοι οι οποίοι εφαρμόζουν, πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Και έχουμε μια ζούγκλα, ένα λαβύρινθο, βαβυλωνίαρη ρυθμίσεων και διατάξεων που δεν γνωρίζουν οι επαγγελματίες τι πρέπει να κάνουν. Και στο κάτω-κάτω δεν γίνεται τίποτα. Ας μην κάνουμε νέες ρυθμίσεις, διατάξεις και ε, ε κανονιστικές ε, διατάξεις ώστε να περιοριστούμε στην εφαρμογή των όσων υπάρχουν σήμερα με έναν ενιαίο εναρμονισμένο τρόπο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υλοποίηση αυτών. Σε σχέση με τους συναδέλφους του ΕΛΚ είχαμε μια ακρόαση που, είχε, που διοργανώθηκε και κάποια πράγματα διαπιστώσαμε. Μας είπαν ομόφωνα οι επιχειρηματίες δεν χρειαζόμαστε πλέον άλλες νέες ρυθμίσεις. Έχουμε καλές και θετικές ρυθμίσεις. Θέλουμε ένα πλαίσιο ενιαίας εφαρμογής και υλοποίησης αυτών των διατάξεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Αναφέρατε ότι η Πολωνία πριν από 7 χρόνια εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα για πρώτη φορά ασκεί την Προεδρία τη. Μπορώ να συναισθανθώ αυτά τα οποία αναφέρατε. Αν μα λέγανε πριν από 20 χρόνια θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα μα λέγανε τρελού. Παλαβούς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ευρώπη έτσι κινηθήκαμε και είναι πολύ καλό αυτό. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στην άσκηση της Προεδρίας από την Πολωνία, διότι ελπίζουμε ότι θα αποβεί προς όφελος όλων στην Ευρώπη. Κάποια πράγματα θα ήθελα να αναφέρω που α, τοποθετηθήκατε κι εσείς επ, ε, αυτών. Στην έκθεση The Grandes Pasquale την προηγούμενη εβδομάδα που εγκρίναμε, συμφωνήσαμε και εκφράσαμε ότι η κατάρτιση για το προσωπικό ασφάλειά σας στα αεροδρόμια πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες, το πιστεύετε αυτό. Και στην Πολωνία και εσείς αυτό κάνετε. Ακριβώς για το προσωπικό ασφάλειας να μην υπάρξει dumping κοινωνικό. Και πώς θα προβείτε, πώς θα προχωρήσετε σε σχέση με αυτά. Αναφερθήκατε στο θέμα των ταχογράφων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές καταχρήσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι και διαφορετική έλεγχη στην Ευρώπη. Είσαστε υπέρ του να είναι αυστηρότερη έλεγχη στην Ευρώπη και μπορείτε με βάση την πείρα σας στην Πολωνία να αναφερθείτε στο πώς μπορεί να γίνει αυτό διότι αναφέρθηκε ότι πήρανε οδηγοί στην αστυνομία και είπανε παρακαλώ σταματήστε με να μην οδηγήσω άλλο γιατί ο επιχειρηματίας ε, το αφεντικό μου με υποχρεώνει και μετά από 14 ώρες να συνεχίζω να οδηγώ σταματήστε με λοιπόν κάντε μου έλεγχο να μην συνεχίσω να οδηγώ Τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν. Έχουμε και τα κοινωνικά θέματα για τις ε, ναυτιλιακές μεταφορές. Έχουμε όμως και οικολογικά θέματα για τη Βαλτική. Αυτά αφορούν όχι μόνο την Πολωνία αλλά και τις όμορες χώρες. Και θα μειωθούν σημαντικά από το 2014 οι εκπομπές ρήπων. Και υποστηρίζεται αυτή την προσπάθεια και την υποστηρίζει η Πολωνία όπως ελπίζω. Μετά αναφέρατε και ένα θέμα τα μεγάλα, τα μείζωνα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις διασυνδέσεις ε, μεταφορών ε, με τις ε, γειτονικέ μας χώρες. Και σε σχέση με τις διασυνδέσεις με τα γειτονικά κράτη τονίστηκε ήδη ότι η διασύνδεση προς τη Λιθουανία και στον άξονα πώς ο βαλτικός σιδηρόδρομος μπορεί να διασυνδεθεί και το πολωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, τα δικά μας διευρωπαϊκά δίκτυα <clears throat> δεν υποφέρουν από το ότι έχουμε λίγα κονδύλια, ισχνά κονδύλια, αλλά χρειαζόμαστε διαφορετική πολιτική. Σε τέσσερα μεγάλα προγράμματα για το τούνελ της Ήραγκα του Μπρένερου το, την σύραγγα ε, Λιών Τουρίνου και ε, άλλα τέτοια μεγάλα προγράμματα αν είχαμε χρηματοδότηση, ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, δεν θα βοηθούσε το να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική όσον αφορά το κλίμα. Χρειάζεται μια, την προστασία του κλίματος, χρειάζεται μια αναθεώρηση αυτής της πολιτικής. Αναθεώρηση. Γνωρίζουμε τον διάδρομο 5, Βία Μπάλτικα, Βασοβία μέχρι τη, Μεσόγειο, μέχρι την Αδριατική. Αυτός ο διάδρομος θα διασυνδεθεί με τον ε, διάδρομο Παρίσι-Μπρατισλάβας. Και η απόφαση στην Βιέννη και το Τώρα θα πρέπει να λυθεί η απόφαση. Θα περάσω από το διάδρομο 5, από την ε, επίπεδη διαδρομή από το Σόπρον και θα μπορέσω με αυτή τη διαδρομή που θα εκμεταλλεύσω με ευρωπαϊκά κονδύλια που θα διευρυνθεί ή θα κάνουμε μια σύραγγα στο Σέμερινγκ στην ε, Αυστρία και να ε, μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο που θα κοστίσει βέβαια πάρα πολλά κονδύλια να μην ε, υλοποιήσουμε άλλα ε, μεγάλα σχέδια αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό. Επί δεκαετίες πολλές φορές ε, ενταφιάζονται, διασπαθίζονται κονδύλια χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Τα λίγα κονδύλια που έχουμε εσείς θα διασφαλίσετε το δυνατόν γοργότερα και πιο αποτελεσματικά θα επεκτείνουν το δίκτυο ώστε να μπορέσει από τις οδικές μεταφορές να μετατεθεί στις σιδηροδρομικές μεταφορές το, ο κυριότερος όγκος εμπορευμάτων. Κάνουμε λόγο για τη δημόσια, την κρατική και την ιδιωτική σύμπραξη. Έχουμε και μια άλλη λύση. Η Ελβετία επειδή δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βρει καλές λύσεις. Μπόρεσε με τα διόδια για τη χρήση των οδικών δικτύων να μπορέσει να κατασκευάσει σύραγγες και υπάρχει ειδικό, ειδικά διόδια για την χρήση των ε, αυτοκινητοδρόμων ε, από πλευρά των φορτηγών οχημάτων. Έχει δείξει η Ελβετία πώ μπορούν να συλλεγούν κονδύλια για τι υποδομέ. Έχουμε την πληροφορία ότι η Πολωνία 1,2 δι ευρώ που προβλεπόντουσαν για το σιδηρόδρομο θα τα μεταθέσει στι χερσαίες μεταφορέ. Έχουμε διαφορετικέ ε, ειδήσει ότι τέλη Ιουνίου έθεσε αυτό το αίτημα λέει η Πολωνία από την άλλη πλευρά ότι επίκειται λέει η διατύπωση αυτού του αιτήματο. Ο Επίτροπος Κάλλας τέθηκε εναντίον και εμεί ως Επιτροπή επίση, διότι αυτό θα ήταν ένα προηγούμενο. Αν γινόταν αυτό, στην πραγματικότητα θα είχαμε πολλά προγράμματα που θα είχαν εγκριθεί για τους σιδηροδρόμους, για τα κράτη-μέλη και θα έλεγαν τα κράτη-μέλη δυστυχώς επειδή δεν τα καταφέραμε θα περάσουν αυτά τα λεφτά από τους σιδηροδρόμους στις χερσαίες μεταφορές γιατί δεν γινότανε. Γι' αυτό θέλω να μου αναφέρετε εσείς τι γίνεται από πλευράς της Πολωνικής Προεδρίας. Να προσέξετε να μην υπάρξουν λανθασμένες προτεραιότητες. Ένα τελευταίο σημείο στα μεγάλα αυτά προγράμματα. <clears throat> Για μένα ήταν ενδιαφέρον σήμερα το πρωί να ακούσω ότι έχετε υπόψη το σιδηροδρομικό σταθμό Lodge που θα μετατραπεί και θα ε, προσαρμοστεί. Έχουμε και σε σχέση με τη Στουτγάρδη αντίστοιχες ε, τέτοιες εμπειρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει ούτε ευρώ γι' αυτό. Η Στουτκάρδη δεν παίρνει δεκάρα γι' αυτό. Στο Μπρουν ήθελαν επίση πάλι να μετατραπεί ένα σιδηρόδρομο, ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν είναι θέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά, η διαμόρφωση σιδηροδρομικών σταθμών. Είναι θέματα των χωρών. Μόνο τι διαδρομέ, τα, τα δίκτυα των διαδρομών χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μετατροπέ σιδηροδρομικών σταθμών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε τις πρώτες πέντε ερωτήσεις και κατόπιν έχω άλλους πέντε αγορητές για το δεύτερο γύρο. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και ιδίως για τις ευχές σας ε, για την Πολωνική Προεδρία. Μας ευχήθηκατε κάθε επιτυχία και κουράγιο και θάρρος. Αλλά θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τις απόψεις σας, οι οποίες ε, αφορούν τα πιο σημαντικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Πολωνική Προεδρία και που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω Ε, τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά το λειτουργικό μπλοκ, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να προκύψει στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Ε, μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό και η Πολωνία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτά τα FABs. Είμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τη Λιθουανία και ελπίζουμε ότι στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας θα υπογραφεί η συμφωνία για την ε, για τον κοινό εναέριο χώρο ε, με στην ε, Βαλτική. Αυτό θα μας επιβεβαιώσει και πόσο σημασία δίνουμε στον ενιαίο ουρανό. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, θα θέλαμε επίσης να εξετάσουμε και την τεχνική διάσταση του ΣΕΖΑΡ. Αυτό το ανέφεραν και ο κύριος Γκρός, αλλά και η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. όσον αφορά τα λοιπά θέματα που σχετίζονται με την αεροπλοεία, όπως για παράδειγμα τους αρωτές σώματος, ε, τους ελέγχους για τα υγρά και τις γέλες, και τα θέματα ασφάλειας ε, στις εναέριες ε, μεταφορές εν γέννη. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα λόγω ζητήματα. Ιδίως το θέμα των σαρωτών. Πρόκειται για ευαίσθητα θέματα, τα οποία άπτονται και των προσωπικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Υπάρχει άλλωστε και το θέμα των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων. Για τους αρωτές ε, υπάρχει κάποια νέα τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την ε, διαβίβαση, τη διάδοση αυτών των νέων τεχνολογιών σάρωσης την περασμένη εβδομάδα στην ε, ε, συνεδρίαση για την πολιτική αεροπορία υιοθετήθηκε μια λύση η οποία ανταποκρίνεται κατά το ίμιση στις απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας των επιβατών και αναφέρεται και σε θέματα ε, σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των επιβατών. Ελπίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει ε, τις νέες ε, λύσεις που προτείνονται για τους αρωτές. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση για θέματα ασφαλείας. Ο κύριος Αλκαντράουι αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν στην ατζέντα του Συμβουλίου πριν από δύο χρόνια. Και τότε, δυστυχώς, ε, τα πράγματα έφτασαν σε αδίέξοδο και σταμάτησε η συζήτηση επί του ζητήματος. Η Πολωνική Προεδρία όμως, ε, στη διάρκεια της προετοιμασίας για την Προεδρία της, ε, ασχολήθηκε με το ζήτημα και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πολιτική βούληση να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση επί του ζητήματος. Δεν γνωρίζουμε βέβαια κατά πόσο θα συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετή συμφωνία ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις ε, για το ζήτημα. Ελπίζουμε όμως ότι στη διάσκεψη που θα οργανώσουμε στη διάρκεια του φθινοπόρου θα μας δοθεί ευκαιρία να ε, συζητήσουμε και το συγκεκριμένο θέμα. τουλάχιστον ε, να ανοίξει μια πλατφόρμα ώστε να επενεξεταστεί το ζήτημα. Για τα TNT τώρα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις ε, μορφές χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε όλες τις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης ε, η βασική βέβαια πηγή είναι ο κρατικός προϋπολογισμός και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αλλά θα πρέπει να αναζητήσουμε με ενεργό τρόπο και νέες μορφές χρηματοδότησης. Ε, γι' αυτό και η Πολωνική Προεδρία σκοπεύει να ξεκινήσει μια συζήτηση για το θέμα αυτό. συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Μεταφορών. Όλοι έχουμε προσωπική πείρα από συμπράξει δημοσίου ιδιωτικό τομέα ως μορφή χρηματοδότησης. Η Πολωνία έχει και καλά και κακά παραδείγματα για τις συγκεκριμένε συμπράξεις. και ε, δεν έχουμε συμπράξεις τέτοιες μόνο για τις κατασκευές αυτοκινητοδρόμων αλλά και για τους σιδηροδρόμους. Και στους σιδηροδρόμους υπάρχουν συμπράξεις ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα για την ε, κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών. Αυτή είναι απάντηση στα όσα μας είπε ο κ. Κράμερ. Και πρόκειται και για καλή εμπειρία διότι δημιουργείται ε, νέα υποδομή. Αλλά φυσικά υπάρχουν και οι αρνητικές πτυχές ε, σε κάποιες περιπτώσεις. Γνωρίζουμε ότι η Eurostat εξετάζει επισταμένα το δημόσιο χρέος, το οποίο ε, προκύπτει από τα συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να μην επιβραδύνουμε τις διαδικασίες και να μην παρακολύσουμε τις ε, κατασκευές ε, υποδομών ε, στα θέματα των μεταφορών ή τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών. Για την ΕΜΣΑ τώρα, τον Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας και το όλο πακέτο για τη θαλάσσια ασφάλεια. Πολωνική Προεδρία ε, το κατατάσσει στις προτεραιότητές της. οι αρχές που διέπουν ε, ε, την ασφάλεια στη θάλασσα ε, θα πρέπει να διέπουν και την κατάρτιση των ναυτικών και αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει απλώς να δημιουργήσουμε μια νέα σύγχρονη αγορά εργασίας, δηλαδή να σταθούμε μόνο στις κοινωνικές πτυχές, αλλά μας ενδιαφέρουν και τα θέματα της ασφάλειας και στη δεδομένη περίπτωση έχει σημασία να μην νομοθετήσουμε υπερβολικά για το συγκεκριμένο τομέα. Και αυτή είναι η θέση που ε, τηρεί το Συμβούλιο. Το σκεπτικό μας είναι ότι δεν θα πρέπει να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία Γι' αυτό ακριβώς ε, γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων ε, της ΕΜΣΑ, η οποία ε, θεωρητικά θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε θέματα ασφαλείας και τις ε, δευτερεύουσες δραστηριότητές της. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Απάντησα νομίζω ε, για τα FABs, τα Functional Space Blocks. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω όσους μου επέστησαν την προσοχή επί του θέματος. Μας ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα το θέμα των σχέσεών μας με τις τρίτες χώρες. Είναι σημαντική αυτή η προσέγγιση για τις μεταφορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και ένα επιπλέον ε, καθήκον σε αυτή την περίπτωση. Ο Πολωνός ε, Πρωθυπουργό, όταν καθόριζε τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας ε, στην, και της παρουσίας στην Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η δημιουργία κατάλληλης εταιρικής σχέσης, ιδίως προς Ανατολάς, είναι ε, μία από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε μια πρακτική επιβεβαίωση της συγκεκριμένη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τον τομέα των μεταφορών. Διότι αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε σχέσεις με τρίτες χώρες και πιο συγκεκριμένα με χώρες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Για τη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, τα πιο σημαντικά ζητήματα που συζητώνται στο Συμβούλιο αφορούν τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση της αγοράς των σιδηροδρόμων, και τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο διαχωρισμός ε, διαχειριστή συστήματος και διαχειριστή υποδομών. Και φυσικά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθοριστεί. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεκινήσει και ένα νέο στάδιο εργασιών, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα και η δέσμη αυτή μέτρων είναι υψής τη σημασίας, διότι οι σιδηροδρομικές μεταφορών, μεταφορές ε, είναι και μεταφορές χαμηλής εκπομπής ε, αερίων. Ε, τίνουμε να το ξεχνάμε, ειδικά σε σύγκριση με τις θαλάσσιες μεταφορές. Ε, αναφέρθηκε και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό όταν ε, αναφερθήκαμε στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά θα πρέπει να το έχουμε και κατά νου όταν συζητάμε τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να ε, εξετάσουμε και τις οδικές μεταφορές, είναι πρόκληση και το ζήτημα αυτό και φυσικά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και αρκετά πράγματα στον τομέα των οδικών μεταφορών. Δεν θα ήθελα να σταθώ σε πάρα πολλά παραδείγματα από την Πολωνία. Στην ε, συζήτηση στην Ολομέλεια έθιξα το ζήτημα και ίσως θα μπορούσα να το πω και εδώ. Από 1η Ιουλίου εφαρμόζουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ε, διοδίων. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά το σύστημα είναι πλέον σε λειτουργία. Γιατί σας αναφέρω το συγκεκριμένο ζήτημα οι τιμολογήσεις υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε το χαμηλότερο τίμημα καταβάλλεται από τους οδηγούς ε, που οδηγούν το πιο καθαρό όχημα, δηλαδή τον οποίων οι κινητήρες παράγουν το χαμηλότερο ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ υγιής τρόπος προσέγγισης του ζητήματος το συζητήσαμε άλλωστε όταν αναφερθήκαμε και στις ευρωβινιέτες, αλλά ε, νομίζω ότι μακρηγορώ σε αυτή την περίπτωση. Ε, το σημειώνω όμως, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα επανέλθω αργότερα. Υπάρχει και το ζήτημα της ε, μεταφορές 1,2 δις ευρώ από τα σιδηροδρομικά στα οδικά ε, στις οδικές μεταφορές. Γιατί έγινε αυτή η αίτηση. Είναι η πρώτη φορά που η Πολωνία εφαρμόζει ε, τόσο μεγάλα προγράμματα υποδομών. Είτε αυτά είναι για το σιδηροδρομικό τομέα, είτε είναι για τον τομέα των αυτοκινητοδρόμων. Και έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια αγορά στην Πολωνία οι ίδιες δυνατότητες της Πολωνίας ε, στον κατασκευαστικό τομέα δεν ήταν επαρκής και γι' αυτό ακριβώς επειδή άλλωστε υπήρχαν και αρκετά σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες ε, ε, επιβράδυναν τις αντίστοιχες κατασκευές στις υποδομές, αρχίσαμε να επιφελούμαστε εμείς από τα αντίστοιχα κοντήλια. Αυτό οδήγησε σε μείωση των τιμών, σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις κόστους ε, που ε, είχαν κάνει οι επενδυτές. Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, βάσει και των αρχών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, ολοκληρωθούν τα προγράμματα αυτά υπό τη συγκεκριμένη προοπτική. Ε, δεν υπάρχουν νέα προγράμματα στο τομέα των σιδηροδρόμων. Ω αρμόδιο υπουργό Μεταφορών δεν θα πρέπει να επιτρέψω μια κατάσταση όπου έστω και ένα ευρώ των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, πηγαίνει χαμένο. Γι' αυτό ακριβώς έγινε η πρόταση να μεταφερθούν αυτά τα κονδύλια στον ε, τομέα των αυτοκινητοδρόμων και στις οδικές υποδομές. Ετοιμάζουμε όμως νέα προγράμματα και στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές αυτή ε, δυσαναλογία, αν θέλετε, θα διορθωθεί και δεν πρόκειται για κάποιο μακρόπνο όραμα. Θεωρούμε απλώς ότι δεν πρέπει να διασπαθιστούν δημόσια κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μεταφορά των κονδυλίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι ίσως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα κονδύλια για μικρότερα προγράμματα, όχι για τόσο μεγάλα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη εξυγχρονισμό κάποιων ε, ε φορτηγών οχημάτων για παράδειγμα. Αυτά όμως τα σκεφτήκαμε αφού ε, σκεφτήκαμε το θέμα της μεταφοράς κονδυλίων. Αν το είχαμε πει νωρίτερα θα είχε αρνηθεί η Επιτροπή. Έχω πανικοβληθεί λίγο, λέει ο Πρόεδρος, γιατί βλέπω ότι περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Δεν μας μένει πολύ χρόνος, δυστυχώς. Θα πρέπει να περιορίσω τους ε, συναδέλφους ε, σε τρία λεπτά. Μετά πρέπει να περιορίσω βέβαια και τον Υπουργό ε, στις απαντήσεις. του κύριο Ζασάντα έχει καταρχάς το λόγο. Θα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας επίσκεψη στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι πολύ που σας συναντούμε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή τύχη, καλή επιτυχία στο έργο σας και συγκεκριμένα σε σχέση με τον νέο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Είστε Πολωνός πολιτικός. Σήμερα θυμίζει η Πολυνέα, θα έλεγα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περιφέρειες που υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν σε αεροδρόμια, αλλά υπάρχουν άλλα μέρη που δεν έχουν ε, ούτε αυτοκινητόδρομους ούτε αεροδρόμια. Υπάρχουν όμως και τοποθεσίες μέρη που δεν έχουν καν βασικές υποδομές, ε, ε, οδικό δίκτυο, εσωτερικές πλωτές οδούς, σιδηροδρόμους. Πρέπει να γίνουν πολλά λοιπόν, γι' αυτό το λέω αυτό. Και πρέπει και εμείς ως χώρα να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα για να εκπληρώσουμε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι για τα νέα χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων τα οποία ε, δημιουργούνται και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες γιατί αυτό θα αποτρέψει και πολλά τροχέα που οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Βελτίωση επίσης περιμένουμε και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη διατροπικότητα ε, των ε, μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται αλλαγές λοιπόν και στα ποτάμια δίκτυα, στο Βιστούλα και ε, σε άλλους ποταμούς στην Πολωνία. Η ασφάλεια λοιπόν, η διατροπικότητα είναι σημαντικές αρχές. Είναι δύο πυλώνες, αν θέλετε, της ε, πολιτικής μεταφορών. Η τρίτη πτυχή, ο πυλώνας, είναι η οικολογία, το περιβάλλον. Και ξέρω ότι στόχος είναι να υπάρχουν πράσινοι διάδρομοι, να είναι οικολογικά τα συστήματα μεταφορών. Αυτός είναι ο στόχος της Πολωνικής Προεδρίας. Πώς στοχεύει να τον υλοποιήσει. Ποια είναι τα σχέδια της Πολωνικής Προεδρίας από αυτού και πώς βλέπετε τις εξελίξεις σε σχέση με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταξύ Βαλτικής και Ανδριατικής. Τι μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένα ε, στο προσεχές εξάμεινο. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα καταρχάς και εγώ να σας καλωσορίσω Έχετε ήδη ακούσει ε, θερμά λόγια από τους προλαλήσαντες, ο κύριος Λιμπεράτσκι. Θέλω όμως να αναφερθώ σε κάτι το οποίο έθιξε ο κύριος Σελκαντράουι. Μιλήσατε για τη στρατηγική σημασία των ευρωπαϊκών δικτύων. Και είναι σημαντικό αυτό. Αλλά ε, έχω δύο θέματα να αναφέρω. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα και τον προπολογισμό, ξέρουμε ότι το Συμβούλιο προτείνει περικοπές της τάξεως ε, ε, του 10% ε, δηλαδή περικοπές κατά 1,02 εκατομμύρια. Σας παρακαλώ αλλάξτε το αυτό κύριε Υπουργέ. Έχει υπάρξει συμφωνία για το θέμα αυτό. Τώρα, 2014-2020. Σε αυτή την περίοδο έχουμε δύο προτάσεις. Αφενός θέλουμε μεγάλη αύξηση ε, των ε, συνδέσμων και των ε, διευρωπαϊκών δικτύων με συνδυασμό δικτύων μεταφορών και διαρθρωτικών ταμείων. Υπάρχουν διάφοροι τομείς από τους οποίους μπορούμε να βρούμε χρήματα. Έχουμε επίσης ε, κάποια σε εκατοντάδες χιλιάδες νέα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, αλλά δεν είναι ομοιόμορφο το σύστημα αυτό. Δεν είναι ένα όλο. Καλό θα ήταν να υπάρχει ολιστική προσέγγιση στην όλη μας στρατηγική. Νομίζω ότι οι Υπουργοί Μεταφορών θα πρέπει να έχουν ε, μεγαλύτερο λόγο στο πώς αυτό θα πρέπει να γίνει. Και ένα τρίτο σχόλιο. Μου άρεσε η προσέγγιση σας σε σχέση με την θαλάσσια οικονομία, σε σχέση και με τις πτυχές της εκπαίδευσης και του κεντρικού ευρωπαϊκού διαδρόμου. Θα μπορούσαμε με τους, βοηθ... τους ε, συναδέλφους από την Τσεχία και την Ουγγαρία να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία και σε σχέση με τον ε, S3 ε, διάδρομο στην πολωνική πλευρά. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή διαδρομή από τις ε, σκανδιναβικές χώρες μέχρι τη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ και προσβλέπουμε στους πέντε μήνες και δύο εβδομάδες συνεργασίας μαζί σας. Κύριος Καντσιάν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Θεωρώ ότι η παρουσίαση που άκουσα από τον Πρωθυπουργό σας στην Ολομέλεια και όσα άκουσα από σας σήμερα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αριστεύσουμε στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Έχετε τη δέουσα ταπεινοφροσύνη και τη δέουσα προετοιμασία. Γι' αυτό λοιπόν σας συγχαίρουμε και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το επόμενο εξάμεινο. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι σε αυτό το εξάμεινο τουλάχιστον όσον αφορά την Επιτροπή μας, έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα. Υπάρχουν τα TNT, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ο ενιαίος ουρανός. Πρόκειται για τους δύο μεγάλους πυλώνες που ε, απαιτούν και περιμένουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Άκουσα τις ερωτήσεις των συναδέλφων μου και τις απαντήσεις σας όσον αφορά τους πόρους και τη χρηματοδότηση. Καλώς το Σεπτέμβριο θα συναντηθείτε με τους υπουργούς και όλα θα είναι εντάξει, αλλά επειδή από τους προκατόχους σας εδώ και δύο χρόνια ακούω πολλές φορές ότι υπάρχει διάθεση για ίδιους πόρους, ε, για project bonds ε, και ούτω καθεξής. Άκουσα δηλαδή τις διάφορες εναλλακτικές ε, ε, περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν ε, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα ήθελα να δεσμευτείτε λίγο περισσότερο σήμερα, να μας πείτε κατά πόσον υπάρχει διάθεση να υλοποιήσετε όσα είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής ε, ο κ. Μπαρόζο και όσα είπε ο Πρωθυπουργό σας σήμερα. Και αν όντω υπάρχει διάθεση, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό του ε, ελάχιστου πόρους που έχουμε τη διάθεσή μας, στη διάθεσή μας, θα τους βάλουμε πάνω σε ένα δοχείο και θα αρχίσουμε να δούμε τι χρηματοδότηση χρειαζόμαστε για ό,τι λείπουν ή θα έχουμε ε, ε, μεμονωμένα προγράμματα χρηματοδότησης για τις μεμονωμένες συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα για τα, ο κάθε κομματάκι υποδομής που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Το ίδιο είναι, μπορούμε να το υλοποιήσουμε όπως θέλουμε. Υπάρχει όμως διάθεση να οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πέρα από την εκλογήκευση και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τα λίγα κονδύλια που έχουμε, ε, επειδή ακριβώς είναι λίγο τα κονδύλια, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε αυτό το άλμα ποιότητας που απαιτείται. Χρειαζόμαστε υποδομές και θα χρειαζόμαστε κατεπηγόντως να παρασύρουμε την οικονομία. Αν η Ευρώπη λοιπόν κάνει αυτή την προσπάθεια, αν εμείς κάνουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τις χώρες μας. Εχθέ έγινε η συζήτηση για την αναδιατύπωση τη δέσμη μέτρων για του σιδηροδρόμους. Ε, το συγκεκριμένο θέμα ε, πάσχει από έλλειψη σαφήνειας. Θέλετε να το οδηγήσετε προ την απελευθέρωση ή θέλετε απλώ να κλείσει το ζήτημα και να ανοίξετε ένα καινούριο ζήτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται κάποιε περισσότερε εγγύσει. Ένα τελευταίο στοιχείο μόνο. Δυστυχώ τρία λεπτά είναι ελάχιστα. Δεν μου φτάνουν από όσα θέλω. Είδα για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, τι ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο προγραμματισμό για τα TEN-T έχετε αφήσει απ' έξω όλα τα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι σωστό αυτό ο προγραμματισμό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι ναι μεν τώρα είναι εκτό Ευρώπη, αλλά για την προοπτική για το 2020 θα πρέπει να δούμε με λίγο διαφορετικό οπτικό πρίσμα όλα όσα ε, πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω ότι είναι λίγα τρία λεπτά, αλλά οι συντονιστέ ε, μακρηγόρησαν λίγο και επομένω ότι ε, τα... Όσοι είναι στον πάγκο πρέπει να μιλήσουν λίγο λιγότερο. Ναι κύριε Υπουργέ και από μένα κάθε ευχή για επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο. Πιο πριν, προηγούμενα, αναφερθήκατε στα θέματα των μεταφορών και είναι ένα καλό παράδειγμα πώς η συνεργασία μεταξύ της Πολωνικής Προεδρίας και της Επιτροπής μας μπορεί να προχωρήσει. Έχουμε άτυπες συζητήσει και στο μέλλον θα τις έχουμε, ώστε να βρούμε ακριβώς στο τέλος των διαβουλεύσεών μας αν έχει νόημα και ουσία σε πρώτη ανάγνωση να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σίγουρα δεν θα ευθύνεται η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή αν καθυστερήσουν τα πράγματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι 25 κράτη-μέλη συμμετέχουν και έχουμε την παράκληση τα έντυπα τα οποία μας αφορούν τα χρειαζόμαστε έγκαιρα. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και για άλλα, όπως για την οδηγία για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση και για το port package, το πακέτο για τα λιμάνια. Είχαμε πριν από κάποια χρόνια εξετάσει και δεν ε, ευδοκίμησε το σχέδιο και τώρα ξαναπερνάει αυτό το θέμα ξανάρχεται θα πρέπει να συζητήσουμε σίγουρα και γι' αυτό και ένα τρίτο τελευταίο σχόλιο και δεν θα χρησιμοποιήσω και τα τρία λεπτά και δεν υπάρχει κάποιο πλήρες ε, ε, πακέτο μέτρων για τα αεροδρόμια. Φυσικά οι υπηρεσίε εδάφου πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, αλλά αν στην φιλελευθεροποίηση προχωρήσουμε μόνο στη ράχη στο σβέρκο των εργαζομένων εις βάρος τους, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό 50 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλέκενστάιν. Ο κύριος Κόχ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Κόχ. Πρόεδρε, ε, κύριε Προεδρεύοντα, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες σας. Κατανοούμε πολύ καλά το πρόγραμμά σας και θα βοηθήσουμε στην υλοποίησή του σίγουρα. Πληροφορίες για τρία θέματα θα ήθελα. Πρώτον, σύντομα, την ανάπτυξη της οικονομίας ε, θέλουμε να την επιτύχουμε στην Ευρώπη. Έχετε μια ιδέα πώς η αύξηση σε σχέση με τις συγκοινωνίες έχει επίπτωση σε αυτό. Δεύτερον, αποδοτικότητα των ενεργειακών πόρων. Όλοι γνωρίζουμε την εξάρτηση των μεταφορών από το πετρέλαιο. Έχετε κάποιες απόψεις για την απαγκίστρωσή μας από τα, το πετρέλαιο. Έχουμε και σε σχέση με τις ε, οδικές μεταφορές ε, σχέδια για την αδειοδότηση, για παράδειγμα, ειδικών ηλεκτρικών φορτηγών για την ε, ε, κυκλοφορία τους υπόρους. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκούρμαϊ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Εδώ βρίσκομαι λέει η κυρία Γκούρμαϊ. Η ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζω ότι θα συνεχίσει το έργο των προηγουμένων προεδριών και θα μπορέσει να συνεχίσει και για την κοινωνική ατζέντα μία από τις προτεραιότητες που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Εσείς αναφέρατε για το εγχείρημα που θα υπάρξει άτυπη ε, συνάντηση των Υπουργών. Θα θέλαμε όμως να γνωρίζουμε ποια θα είναι η κύρια, τα κύρια θέματα και τα σχέδια που έχετε για την περιφερειακή συνιστόσα των μεταφορών και πώς σε σχέση με τις υποδομές θα υπάρξει ανάπτυξή τους σε σχέση με τις διαφορετικές περιφέρειες και για την χρηματοδότηση. Φυσικά πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα ε, σχέδια για τη νέα πολιτική συνοχή. Πώς εντάσσονται όλα αυτά στο πρόγραμμά σας μετά σε σχέση με την ανατολική γυτνίαση, την ανατολική γειτονική σχέση. ποιε είναι οι προτάσεις σας σε σχέση με την ανατολική γειτονική σχέση και τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτές τις χώρες που θα πρέπει να έχουμε διασύνδεση με αυτές. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω την κοινωνική διάσταση του συνολικού τομέα των μεταφορών και πρέπει εδώ να δούμε την ε, διάσταση αυτών των κοινωνικών θεμάτων και θα ήθελα να υπογραμμίσω το θέμα των ε, υπηρεσιών και το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών τι προγραμματίζει να κάνει στις εναέριες μεταφορές με τις φθηνές εταιρείε φθηνών ναύλων η Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστώ. Νίχτενμπεργκερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα. Θα ήθελα κάποια θέματα να αναφέρω που πιο πριν τα θίξατε εσείς. Το ένα αφορά τα προγράμματα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια διαπιστώνει ότι σε μεγάλα τέτοια σχέδια λόγω της μεγάλης διάρκειας προκήρυξης υπάρχουν δυσκολίες αλλά και σε μικρότερα προγράμματα πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι και εκείνοι που πήραν καλά σε ε, βραβεία ή ε, είχαν επιδόσεις, ε, στο τέλος τέλος είχαν προβλήματα. Αυτός αυτό το πρόβλημα, αυτός ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται. Και θυμάμαι δεν ήταν ένα θέμα ΠΠΠ, αλλά είχαμε σε σχέση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ε, πίεση που ε, υπήρξε ώστε υπό την ε, φθηνότερη τιμή προσφοράσα πήρανε κάποιοι Κινέζοι ε, μια δουλειά. Νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της ε, φθηνής ανάθεσης ή της ε, φθηνότερης προσφοράς ε, να τύχει ιδιαίτερη προσοχή από πλευρά σας και σε σχέση με ένα άλλο πακέτο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο σε περίοδους κρίσης ε, όπου εμείς, ας το πω με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι οι χώρες αποτυγχάνουν στη χρηματοδότηση. Ακόμα και αν υπάρξει διπλασιασμός ε, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη που λόγω περιορισμών και ε, ασφυξίας οικονομικής δεν μπορούν να δράσουν. Αλλά αν υπάρξει μετάθεση μόνο προς την μετάθεση υπέρ του φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα πρέπει να δράσουμε να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην περίοδο αυτής της κρίσης, σε αυτή τη συγκεκριμένη κρίση, πρέπει να αναθεωρήσουμε την λογική που μας εμπνέει, να ξεφύγουμε από τα μεγάλα πομπόδι ε, προγράμματα και να ε, μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σε ένα εφικτό πλαίσιο δυνατότητες ενεργοποίησης από πλευράς μας. Για το ground handling, τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια, παρακαλώ να προσέξουμε να μην υπάρχει συνέχιση διαρκώς της αρχής της ιδιωτικοποίησης και να ξεπεράσουμε το νόημα του αποτελεσματικού ή ρεαλιστικού διότι έχουμε φτάσει πια τόσο μακριά έχουμε μεταθέσει τα πράγματα τόσο που η επικοινωνία η συνάφεια χάνεται και ο χαμένος πάντα σε αυτό το παιχνίδι είναι ο επιβάτης, είναι οι επιβάτες μπορώ δυστυχώς και από την ίδια μου την πείρα να το αναφέρω αυτό, ευχαριστώ σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ ο συνάδελφός σας θα περιμένει πρώτον θυρών. Αν μπορείτε όμως εσείς σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται να απαντήσετε, θα είμαστε ευγνώμονες. Παρακαλώ Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να αυτοπιθαρχήσω και να είμαι πραγματικά πολύ σύντομος στις ερωτήσεις που μου διατυπώθηκαν. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λέγοντας για τον αναφερόμενο στον ενιαίο ευρωπαϊκό θέρα. Το ανέφερα στην προηγούμενη μου παρατήρηση για τους ε, ευρωπαϊκούς ουρανούς. Δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα. Γι' αυτό θα αναφερθώ στη δεύτερη ερώτηση για τους πράσινους διαδρόμους στους οποίους αναφερθήκατε. Η Πολωνική Προεδρία θα κάνει κάθε προσπάθεια και σίγουρα θα ασχοληθεί με την δημιουργία αυτών των πράσινων διαδρόμων. Πρέπει όμως καταρχήν πρώτα να συμφωνήσουμε και να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ορισμός, ένας σαφής συγκεκριμένος προσδιορισμός του TST πράσινος διάδρομος, διότι δεν υπάρχει ένας τέτοιος γενικά αποδεκτός δόκιμος ε, προσδιορισμός που να γίνεται δεκτός από όλους. Πρόκειται για διαδρόμους της ε, διατροπικής μεταφοράς με διαφορετικά μέσα και φορείς μεταφορών και για την μείωση των εκπομπών ρήπων φυσικά που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αυτό είναι το νόημα αυτών των πράσινων διαδρόμων. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως την εργασία μας να αποσαφινιστούν τα πράγματα στο Σεπτέμβριο. Στο Σετσίν θα δημιουργηθεί μια ευρύτερη τέτοια ακρόαση, μια τέτοια συνάντηση. Όλοι αναμένουμε από τη συνάντηση στο Σετσίν να συζητηθεί το θέμα και να εξεταστεί το θέμα των πράσινων διαδρόμων. Τώρα, τι έχουμε εδώ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσα να προσθέσω και να πω ότι ο κέντρο ευρωπαϊκός διάδρομος φυσικά είναι σημαντικός και φυσικά υλοποιεί ε, τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σίγουρα. Όμως, στο Σκετσίν θα πρέπει να συζητήσουμε, στην Πολωνία για αυτά τα πράγματα, όταν έρθει η ώρα εκείνη. Και για τον Ευρωβουλευτή κύριο Λιμπεράτσκι, μου έθεσε ένα πολύ δύσκολο, δυσχερέστατο ερώτημα. Διότι είναι το δυσκολότερο θέμα να συζητήσει και να διαπραγματευτεί κανείς για τα χρήματα, τα κονδύλια. Όταν κάνουμε λόγο για τα κονδύλια, για τον προϋπολογισμό, ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε και υπέβαλε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού. Και μάλιστα στις 29 Ιουνίου. Τώρα εμείς θα πρέπει να αναμείνουμε τις λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα δημοσιονομικά πλαίσια και προγράμματα και δημοσιονομικά πλαίσια και θα πρέπει να δούμε μέσα στο πολιετές αυτό πλαίσιο αν θα υπάρξουν επαρκή κονδύλια για τις υποδομές ιδιαίτερα για φιλοπεριβαλλοντικές υποδομές. Ελπίζω, ευελπιστώ ότι αυτό θα είναι εφικτό, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλά θα εξαρτηθούν και από την δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι. Είμαι πεισμένος ότι από κοινού εμείς, κυρίες και κύριοι, εδώ θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να τα επιλύσουμε όσο το καλύτερο γίνεται και σε αυτόν τον τομέα επίσης. Τώρα, στην συνέχεια κάτι άλλο. Τα οικονομικά θέματα και από τον κύριο Κάντσαν προαναφέρθηκαν στην παρέμβασή του. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και να αναφέρω πάλι αυτό το οποίο προανέφερα. Πρέπει να αναμείνουμε μέχρι ότου να έχουμε το εξειδικευμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα κονδύλια για τον προϋπολογισμό. Και μόνο τότε θα μπορέσουμε, τότε θα είναι δυνατόν εξειδικευμένα να τοποθετηθούμε από αυτών των προτάσεων και αν θα είναι αναγκαίο θα, τότε θα πρέπει από κοινού να αναλάβουμε να πρωτοβουλίες και μέτρα και κάποιες αποφάσεις. Και στη συνέχεια ε, ακολουθεί ε, και, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάρμοδη. Τώρα για το πακέτο μέτρων για, τον, για τους σιδηροδρόμους υπήρξε ερώτηση και για αυτό το θέμα. θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα θέματα που αφορούν αυτό το χαρτοφυλάκιο με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση, την επανεξέταση, επανεκπώνηση του πακέτου για τους σιδηροδρόμους και με αφορμή αυτό ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τώρα προς τον κύριο Φλέκενστάιν. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Εσείς αναφερθήκατε σε θέματα που αφορούν το πακέτο για τα αεροδρόμια. Για μας αυτό το πακέτο για τα αεροδρόμια είναι μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες της ε, πολωνικής μας προεδρίας όσον αφορά τον τομέα των θεμάτων μεταφορών. Και εδώ θα επικεντρωθούμε ακριβώς σε εκείνα τα θέματα και ζητήματα που αφορούν τις εδάφιες υπηρεσίες, υπηρεσίες εδάφου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε τις άλλες πτυχές ε, σε σχέση με τα αεροδρόμια, ε, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά παρόλα αυτά το πιο σημαντικό είναι να σημειωθούν πρόοδοι στον τομέα των υπηρεσιών ε, εξυπηρέτησης εδάφους και διεκπαιρέωσης στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι κάπως πρόημο να επισέθω σε λεπτομέρειες, διότι τα έγγραφα δεν τα έχει ακόμα δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν τα έχει ακόμα καταθέσει, δεν βρίσκονται επί τραπέζης. Λαμβάνουμε υπόψη πόσο μεγάλη σπουδαιότητα δίνεται σε αυτό το θέμα κύριε Ευρωβουλευτά και σίγουρα θα σημειώσουμε και θα λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα στην εξέταση που θα τύχει στο μέλλον. Και σίγουρα θα ισχύσει αυτό και το οποίο ανέφερε και η κυρία Γκούρμαϊ στη δική της παρέμβαση. Εξίσου λαμβάνεται και αυτό υπόψη. Νομίζω απάντησα σε σχεδόν όλες σας τις παρεμβάσεις και παρατηρήσεις. Θα ήθελα γενικότερα τώρα, σε ένα γενικότερο πνεύμα και πλαίσιο, να τοποθετηθώ σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια επιρροή ασκεί η ίδια η Λευκή Βίβλο στο Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιες συνέπειες υπάρχουν. Στόχος μας είναι και πρέπει να είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τις μεταφορές με ενιαίο εναρμονισμένο τρόπο. Πρέπει να μεριμνήσουμε αυτό το κοινοτικό, κοινό ενιαίο πλαίσιο να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό. Και γι' αυτό θα πρέπει τα αντίστοιχα μέσα και εργαλεία να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Μέσα σε αυτά ανήκουν και τα χρηματοοικονομικά μέσα ή εργαλεία. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο μύτος της Αριάδνης, η εργαλεια και αυτο θα πρεπει να ειναι ο μυτος της Αριάννης η πορεια που θα ακολουθήσουμε ως Προεδρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Προεδρία που απαντήσατε στα ερωτήματα των ε, βουλευτών. Δυστυχώ ξέρω ότι υπήρχαν και συνάλφοι που ήθελαν έστω και τελευταίες να θέσουν τις ερωτήσεις τους, αλλά δυστυχώ περιμένει υπομονετικά έξω από την αίθουσα υπουργό ε, Τουρισμού και γι' αυτό δυστυχώ πρέπει, επειδή είναι ε, περασμένη ώρα, γύρω στα 4.30 είχαμε πει, και εγώ ήθελα να κάνω ερωτήσεις και εγώ αναγκάστηκα να μην μιλήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ πάντως. Καλή επιτυχία. Ο υπουργό, αν έχει Ο Υπουργός Ομπιαράς την καλοσύνη να έλθει εδώ στο Δήμο. please. Those people who are not here to listen to the minister. Όσοι δεν ε, θέλουν να ακούσουν την Υπουργό, ας συζητήσουν, κάνουν τα παιδαγάκια τους εκτός. Εκτούς παρακαλώ. So that those of us who do want to listen to... minister... Όσοι θέλουν να ακούσουν την Υπουργό, και η οποία θα μας ε, διαγραφήσει το πρόγραμμα της Πολωνικής πρόεδρες για τον τουρισμό μπορούν ε, με ησυχία να ακούσουν την Υπουργό. Καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Καθυστερήσαμε γύρω στα 5-6 λεπτά. Τώρα που έφυγε ο Υπουργό Μεταφόρων μπορώ να τον κατηγορήσω γιατί δεν είναι εδώ για να περασπιστεί τον εαυτό του, αλλά τέλο πάντων. Εσείς λοιπόν εκπροσωπείτε την Πολωνική Προεδρία στο τομέα του τουρισμού. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά το ότι μπορώ σήμερα να σας προσφωνήσω στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών και να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας όσον αφορά τον τουρισμό ακριβώς. Και κατανοώ και γνωρίζω ότι τα θέματα μεταφορών είναι εξαιρετικά σημαντικά φυσικά και για τον τουρισμό είναι προϋπόθεση το θέμα των μεταφορών. Γι' αυτό <clears throat> πρέπει να τονίσουμε και αυτή την πτυχή. Κυρίες και κύριοι, αν επιτρέπετε τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε σημαντικά θέματα που άπτονται του τουρισμού. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα πόσο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τόν τον σημαντικό οικονομικό τομέα τον σημαντικό οικονομικό τομέα τον υποστηρίζει και εσείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Πολωνική Προεδρία και εγώ προσωπικά πλήρως εμπλεκόμεθα και δεσμευόμεθα Δεσμευόμαστε για μια συνέχιση αυτής της καλής συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου αυτή η καλή θετική συνεργασία ήδη κατέστησε εφικτό σημαντικέ πρόοδοι να επιτευχθούν όσον αφορά την πολιτική για τον τουρισμό, ιδιαίτερα μετά την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Και θα έλεγα σε αυτόν τον κύκλο ενώπιον των μελών, μπορώ να πω ότι όλοι γνωρίζουμε φυσικά πόσο σημαντικό είναι ο τομέα του τουρισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα οικονομικός που έχει μεγάλη επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση και οδηγεί η εικόνα της Ευρώπης παγκόσμια να βελτιώνεται και ο πολιτισμικός μας πλούτος, ο πολυσχηδής χαρακτήρας των πολιτιστικών θεμάτων να μπορούν να δίνουν μια εξαιρετική εικόνα. 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και προσφέρουν απασχόληση. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι συνολικά περίπου 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 4% των, των εργαζομένων εργάζεται στον τομέα του τουρισμού. Στο ευρύτερο πλαίσιο θα μπορούσε κανείς να πει ευρύτερα ότι δημιουργείται 10% του ΑΕΠ και 11%, 10 ε, της απασχόλησης και 11% των ε, θέσεων απασχόλησης όσον αφορά το ΑΕΠ. Και στον παγκόσμιο ανταγωνιστικό και στην ανταγωνιστικότητα έχει ιδιαίτερη αξία ο τουρισμός. Είμαστε ιδιαίτερη επιλογή ως χώρες προορισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την οικονομική κρίση και τα πλήγματα που υποστήκαμε ο τουρισμός, ο τομέας στον τουρισμό πραγματικά μπορώ να πω ότι πουλώνονται οι πληγές και ανακάμπτει. Υπάρχουν όμως και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός ευρύτερα. Και για το σύνολο του τουριστικού τομέα προσφέρονται όμως και ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες. Αυτές οι νέες δυνατότητες είναι εκείνο που πρέπει να αναλυθεί εδώ. Εδώ χρειαζόμαστε εντατικές δραστηριότητες που θα οδηγήσουν ο τομέας του τουρισμού να ανακάμψει και να βελτιώσει την θέση του παγκόσμια και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Η συνθήκη Λισαβόνας διευρύνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον τουρισμό. Αν δούμε το άρθρο 6 της συνθήκης, τώρα έχει πλέον αρμοδιότητες χειροπιαστές η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες να υποστηρίξει, να συντονίσει, να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών μελών. Σε καμιά περίπτωση όμως ε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει, να υποκαταστήσει τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Είναι λοιπόν ε, η ενίσχυση του ανταγωνισμού σε πρώτο πλαίσιο, σε πρώτο επίπεδο, η τόνωση του τομέα του τουρισμού Πάντα έχοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη ε, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνδυάζεται στενά με την αηφορία, με την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτός ο στόχος ε, σαφέστατα αναφέρεται στην οικονομική στρατηγική και στους στόχους για το 2020 στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα για την οικονομία μας και την πολιτική μας όσον αφορά αυτούς τους στόχους, ο τουρισμός διαδραματίζει σίγουρα έναν ξεχωριστό ιδιαίτερο ρόλο. Αν δούμε αυτές τις προτεραιότητες στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, μπορεί κανείς να πει ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε μια ανακοίνωση πέρυσι ώστε η Ευρώπη να γίνει το σημαντικότερο, τουριστικό σημαντικότερος τουριστικός στόχος παγκόσμια και να δημιουργηθεί ένας, ένα νέο πλαίσιο τουριστικό από πλευράς της Ευρώπης. Σε αυτή την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ανακοίνωση δείχνει τη σωστή κατεύθυνση, του σωστού προσανατολισμού. πώς μπορεί να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Τέσσερις άξονες αναφέρονται για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, αηφορία στην ανάπτυξη, προώθηση και προαγωγή της Ευρώπης ω σημαντικότερου στόχου του τουριστικού στόχου και η βέλτιστη χρήση των και εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μηχανισμών για τον τουρισμό. Σε αυτές τις τέσσερις προτεραιότητες ως άξονες έχουμε και τη στρατηγική του 2020 που ε, ταιριάζει και προσαρμόζονται αυτές οι προτεραιότητες σε αυτούς τους στόχους. Οι προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται καταρχήν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Ανάλυση και αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, συστάσεις, συμπεράσματα. Αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τώρα στη σημερινή συγκυρία δύο χρόνια μετά την έκρηξη της κρίσης και μετά την έκρηξη και του ηφαιστείου που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στον τουριστικό τομέα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Μετά από αυτά τα γεγονότα που σημειώθηκαν επίσης και στη Βόρεια Αφρική από την άλλη πλευρά πρέπει να εξεύρουμε νέες κατευθύνσεις για τον τομέα του τουρισμού και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε. Τώρα από την άλλη πλευρά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Για την ανταγωνιστικότητα η Πολωνική Προεδρία θα ήθελε η συζήτηση να επικεντρωθεί και να δομηθεί σε τρεις άξονες. Διεύρυνση των κοινωνικών οικονομικών θεμελίων και για τον κοινωνικό τουρισμό. Θέλουμε το επιχειρήν, το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προαχθεί, να υπάρξουν οι αναγκαίε προσαρμογές και οι αναγκαίε καινοτομές όσον αφορά την διεύρυνση των οικονομικών κοινωνικών ε, βάσεων και δεδομένων. Θέλουμε να υπάρξει ένας καλύτερος ορισμός και συντονισμός των στοιχείων και δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Και αυτά τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και να κλείσουμε, να καλύψουμε τα κενά και τα χάσματα. Είναι σημαντικό όχι μόνο να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία, χρειαζόμαστε και καλύτερη στατιστική, καλύτερα στατιστικά στοιχεία που να χρησιμοποιούν την ίδια στατιστική βάση και να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Και επιπλέον θεωρούμε ότι η η κάλυψη από πλευράς πληροφοριών μέσα σε στενή συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να διεξάγεται και να συλλέγονται αυτά τα στοιχεία ιδιαίτερα όσον αφορά δημογραφικά θέματα και θέματα κλιματικών αλλαγών, διαφορές όσον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά και γεγονότα συμβάντα όπως την έκρηξη αυτού του ηφαιστείου. Εδώ αυτά είναι σημαντικά, εδώ πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν τις σωστές απαντήσεις στις νέες ανάγκες που απορρέουν και τίθενται από μια δεύτερη κατεύθυνση αυτών των, αρμο... των δραστηριοτήτων μας κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας ο Σάξονας θα είναι καινοτομίε και νέες ε, τεχνολογίες και, ε, και τεχνολογία στις, στην πληροφόρηση και τις πληροφορίες. Πολύ σημαντικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την ενδυνάμωση του τουριστικού τομέα και τη διασύνδεσή του με άλλους οικονομικούς τομείς δραστηριο, δραστηριοτήτων. Η εκμετάλλευση πληροφοριών, δεδομένων και τεχνολογιών επικοινωνίας είναι σήμερα τελείως διαφορετική από κράτος σε κράτος και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Εξαρτάται από την κατάτηση, το επίπεδο κατάτησης και την χρηματοδότηση σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Πολλές φορές ε, απουσιάζει η αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να προσαρμοστούν όπως πρέπει σωστά αυτές οι επιχειρήσεις ή να εκμεταλλευτούν σωστά τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τα κενά, τις που υπάρχουν και να βοηθήσουμε να καλυφθούν. Οι νέες τεχνολογίες σε κάποιους τομείς ε, ήδη έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω το να είναι κανείς ε, αποτελεσματικός είναι σημαντική υπόθεση και εδώ πρέπει να σημειωθούν πρόοδοι συνειλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων θα ήθελε η Πολωνική Προεδρία να επικεντρωθεί στο εξή. Να υπάρξει ένα φόρουμ για τον τουρισμό στην Ευρώπη που θα διοργανωθεί από τις 5, ε, από τις 5 Οκτωβρίου στις 7 Οκτωβρίου στην Κρακοβία. Ένα σημαντικό φόρουμ, ένα βήμα για τους εκπροσώπους του τουρισμού και τους εκπροσώπους των διοικήσεων και κρατικών αρχών που από πλευράς κρατών μελών είναι συναρμόδιες και συναρμόδια άτομα εδώ τα πιο σημαντικά θέματα θα πρέπει να μπορέσουν να εξεταστούν όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με αυτό το φόρουμ για τον τουρισμό θα έχουμε μια άτυπη σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο θέμα θα είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας απασχολήσει και οι τρόποι υλοποίησης και εφαρμογής όσον αφορά τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την ε, πολιτική για τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Ιούνιο του 1910. Ελπίζουμε ότι αυτή η Υπουργική Σύνοδος θα είναι αποτελεσματική και θα δώσει τη δυνατότητα να γνωστοποιηθούν τα μέτρα και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει αξιολόγηση ή να υπάρξει η αναγκαία τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών των μέτρων και προτάσεων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Θέλω να προσθέσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη επανειλημμένα κατέδειξε στο παρελθόν ότι για σας τους Ευρωβουλευτές ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας. Πολλές δραστηριότητες προωθήθηκαν μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, τα προκαταρκτικά μέτρα όσον αφορά το πρόγραμμα Καλυψό. Εδώ για παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό επίσης και η αύξηση της απασχόλησης και η εξισορρόπηση όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την απασχόληση στον τομέα του τουρισμού. Αυτές οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σημαντικές και είχαν ε, θετικές επιπτώσεις στις τουριστικές δραστηριότητες και έδωσαν νέα όθηση όσον αφορά τις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις συνθήκες της Λισαβόνας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Ευρωβουλευτές της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις μεταφορές και τον τουρισμό, για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για την ανάπτυξη ενός τόσο σημαντικού οικονομικού οικονομικού συντελεστή στην Ευρώπη όπως του τουρισμού. Έχω θετική πολιτική και εμπειρία σε σχέση με τη συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Ελπίζω ότι το πολωνικό πρόγραμμα της Προεδρίας που μπόρεσα να σας παρουσιάσω εξ ονόματος της Πολωνικής Προεδρίας σας ικανοποιεί. με στη διάθεσή σας για περαιτέρω αποσαφηνήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πέντε είναι οι ομιλητές προς το παρόν. Μπορώ να κλείσω τον κατάλογο. Ξεκινούμε με τον κύριο Φιντάντς από το ΕΛΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Καταρχάς ε, ασπάζομαι και δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση κάποιες από τις προθέσεις της ε, Πολωνικής Προεδρίας ε, που θέλατε να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας για το εξάμεινο. Κάποια τα βρήκα ε, πολύ σημαντικά. Έξι μήνες είναι λίγοι μεν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες ε, στα θέματα της εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων για τον τουρισμό, διότι υπάρχει μια κοινή πολιτική βούληση μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε και μια ανακοίνωση η οποία πλέον υλοποιείται με συγκεκριμένε δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει το Σεπτέμβριο την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, που είναι ένα δεύτερο σημαντικό πέρασμα για την ενίσχυση της στρατηγικής για τον τουρισμό. Είχαμε και μία έξοχη σχέση με τις προηγούμενες προεδρίες, ιδίω με την Βελγική Προεδρία, η οποία ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Οκτωβρίου πέρσι ε, έδωσε μια ιδιαίτερη όθηση στα θέματα του τουρισμού. Επομένως υπάρχει ένα δυνητικά θετικό πλαίσιο το οποίο ελπίζω η Προεδρία σας να αυξήσει. Ξεκινώ με το θέμα των πόρων απευθείας. Διότι όπως γνωρίζουμε, οι πόροι που προβλέπονται στον προπολογισμό του 2012 για τον τουρισμό είναι ελάχιστοι, ε, όπως άλλωστε γίνεται πάντα. Ε, το είπαμε άλλωστε και στην έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2012 στην ε, σχετική μας γνωμοδότηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ε, για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 υπάρχει ένα άνοιγμα, ε, όχι τόσο για να αποκτήσουμε όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένως συγκεκριμένε γραμμές προϋπολογισμού για τον τουρισμό, διότι αυτό είναι απαραίτητο και σημαντικό και είναι σημαντικό να προβλέψουμε και πόρους για τον τουρισμό στα πλαίσια του προγράμματος για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αλλά για να ε, δώσουμε κίνητρο στα κράτη-μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο τμήμα των, χρη... κονδυλίων που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Υπάρχουν κονδύλια τα οποία πολλές συχνές πολύ συχνά μένουν κρυφά και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και καλό θα ήταν να γίνεται μια καλύτερη χρήση αυτών των κονδυλίων. Υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Στο πρόγραμμά σας γίνεται μια σημαντική έκκληση ως προς την ανάγκη να επενεξετάσουμε την οδηγία για τα all-inclusive ταξίδια. Εσείς ε, αναφερθήκατε και στο επεισόδιο των εκρήξεων του ηφαιστείου γεγονότα τα οποία ε, μαζί με τα όσα είχαμε στην ε, αραβική ε, περιοχή αυτή την άνοιξη οδήγησαν σε αλλαγές και θα πρέπει να υπάρχει σύντομα ένα κείμενο, άλλωστε το Κοινοβούλιο το ζητάει ε, επισταμένα εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει και ένα ακόμα σημαντικό θέμα το οποίο αφορά την ποιότητα των τουριστικών μας προσφορών. Εμείς αποφασίσαμε να πιστέψουμε σε μια ευρωπαϊκή ε, στρατηγική για τον τουρισμό επειδή σήμερα η αγορά είναι πολύ πιο μεγάλη, μπορούμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή ε, Επικράτεια πολλούς τουρίστες από άλλες υπήρους και επομένως θεωρούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να νικήσει σε αυτή την ε, πρόκληση εάν επενδύσει σε υπηρεσίες ποιότητας. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη και με τους αρμόδιους του τομέα για να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε ήδη αναπτύξει στο παρελθόν ε, ως προς, τις, ε, ως προς την ποιότητα κάποιων χωρών και σας ζητούμε να ενισχύσετε τα θέματα αυτά διότι μόνο αν αναπτύξουμε την ποιότητά μας μπορούμε να νικήσουμε σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση. Υπάρχουν ε, και κάποια ζητήματα που αφορούν τις αναδιόμενες χώρες οι οποίες δεν είναι πλέον αναδεόμενες αλλά είναι πραγματικότητα. Το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίων. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι αποκλειστική δική σας αρμοδιότητα, αλλά επικαλύπτεται και με τις αρμοδιότητες των Υπουργών Εσωτερικών, των Υπουργών Δικαιοσύνης και των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμείς καθημερινά ε, βλέπουμε πως το ένομο δικαίωμα των κρατών μελών να προσπίσουν τα σύνορά τους και να ρυθμίσουν ε, ε, την είσοδο στη χώρα τους γίνονται για τις συγκεκριμένες χώρες ένας περιορισμός από πλευράς ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές διαφορές ε, στα χρονικά όρια και στον τρόπο έκδοσης των συγκεκριμένων θεωρήσεων και αυτό φυσικά δυσχεραίνει τις τουριστικές μας επιχειρήσεις. Μια τελευταία παρατήρηση. Θεωρώ θετικές κάποιες από τις προτεραιότητες που ανακοινώσατε. Το ICT είναι θεμελιώδου σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αναπτύσσει μια δράση επί του θέματο. Εμεί πρέπει να την υποστηρίξουμε με Σθένου. Θα πρέπει να υπάρχουν μικροεπιχειρήσει και μεσέ επιχειρήσει που θα έχουν πλατφόρμε πληροφορική με χαμηλό κόστο για να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα ε, και την ε, προβολή των επιχειρήσεων αυτών στο διαδίκτυο. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα και της επιμόρφωσης. Μια επιμόρφωση η οποία δεν θα είναι πλέον απλώς και μόνο κατάρτιση του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με την πελατεία, του μάγειρα, του ξενοδόχου ή του εστιατόρα, αλλά θα είναι και μια επιμόρφωση που θα έχει στόχο ε, να προσελκύσει ροές τουριστών από τις άλλες υπήρους. Είναι σημαντικό διότι ακόμα και σήμερα υπάρχει υπάρχει μια πολύ σημαντική ε, τουριστική διάσταση που επικεντρώνεται στην εσωτερική αγορά. Το μεγαλύτερο τμήμα των Ευρωπαίων τουριστών είναι Ευρωπαίοι από άλλες χώρες, επομένως θα πρέπει να προσελκύσουμε και τις αγορές από τις άλλες υπήρους και θα πρέπει να κάνουμε κάτι προς αυτή την ε, ε, κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, καλή δουλειά και θα τα πούμε στην Κρακοβία. Ευχαριστώ κύριο Δανέλης από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσία σας εδώ και για αυτά που μας είπατε. Ως γνωστό, ο τουρισμός ε, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα νηπιακά του βήματα ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ότι ο τουρισμός πρέπει να είναι κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και αν θα ήταν δυνατόν να μας πείτε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχετε σκοπό να πάρετε ε, και σε ποια συγκεκριμένα ζητήματα ώστε να αντιληφθούμε ότι πρέπει να χαράξουμε κοινή στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ε, δεύτερο, θα ήθελα να επισημάνω μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ενώ όλοι συμφωνούμε ότι ο τουρισμός είναι μία από τις βασικές ε, πηγές εισοδήματος αλλά και θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι ιδιαίτερα σε αυτήν τη συγκυρία οικονομικής κρίσης ε, στον τουρισμό έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες για να ανακάμψουν τοπικές κοινωνίες και τοπικές οικονομίες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία πρόβλεψη ή σχεδόν καμία ε, στον προϋπολογισμό μας αυτής της δημοσιονομικής περίοδου αλλά δυστυχώς και του επόμενου πολιετούς πλαισίου ε, ικανή να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές και τα θεσμικά μέτρα τα οποία φιλοδοξούμε να πάρουμε σε αυτήν την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα να μου πείτε εάν σκοπεύετε να πάρετε πρωτοβουλίες προς το Συμβούλιο αλλά και προς την Επιτροπή για να αρθεί αυτή η μεγάλη αντίφαση. Και τέλος, πολύ σύντομα, θα σταθώ σε δύο από τα θέματα που ο συνάδελφος Φιντάντσα ανέφερε, γιατί θεωρώ ότι είναι κομβική σημασίας. Πρώτο, αν σκοπεύετε να πάρετε κάποια ε, πρωτοβουλία για τη ρύθμιση επιτέλους του All Inclusive, για την άρση πολλών στρεβλώσεων και προβλημάτων που δημιουργεί και στον οικονομικό ανταγωνισμό, αλλά και προβλημάτων που θέτει σε κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό ε, επίπεδο στις περιοχές που αυτός αναπτύσσεται. Και δεύτερο, αν σκοπεύετε να πάρετε πρωτοβουλία στην ε, διευκόλυνση ε, της έκδοσης των τουριστικών ε, βίζας, κυρίως από τις χώρες BRIC, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, κυρία Υπουργέ. Και προσωπικά σε εσά αλλά και στο σύνολο της Πολωνικής Προεδρίας σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί όλοι θα επωφεληθούμε από αυτό. Μιλήσατε για το βιώσιμο τουρισμό, όλοι θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί ο τουρισμός. Είπατε για αυτό το φόρουμ ε, του τουρισμού στην Κρακοβία. Θα ήθελα να μας πείτε για ποιο θέμα θα είναι. Ήδη στη Μαντρή είχαμε συζητήσει τα πολιτισμικά, ε, τις πολιτισμικές δεξιότητες τότε στη Μαδρίτη. Τώρα λοιπόν γιατί θα μιλήσουμε. Επίση, ό,τι αφορά το βιώσιμο τουρισμό, ο τουρισμός ε, με ποδήλατο, με δίκυκλο, επίσης είναι σημαντικός ε, και έχει δεσμευτεί η Κομισιό να έχουμε του ευρωπαϊκούς ποδηλατοδρόμους. Εσείς ε, θα δεσμευτείτε προ αυτή την κατεύθυνση και αν ναι, πώ θα στηρίξετε αυτές τις υποδομές. Σηματοδότηση για αυτούς τους διαδρόμου ποδηλατών κτλ. Και να είναι πρότυπο για άλλε χώρε αυτό. Σημαντικό και αυτό το στοιχείο έχουμε και το πρωτόκολλο για τον τουρισμό σε σχέση με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί. Τι γίνεται σε σχέση με αυτό το πρωτόκολλο, πώς θα το ενδυναμώσετε και πώς θα εφαρμοστεί. Και κυρίως όταν πρόκειται για τις μεγάλες προσφορές low cost και all inclusive, χαμηλού κόστους και συμπεριλαμβανομένων όλων των παροχών θα πρέπει να εξεταστεί αυτή η πτυχή. Η αηφορία στον τουρισμό δίνει μεγάλες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε διασύνδεση μεταξύ αηφορίας και οικονομικού προτερήματος για τους μικρούς, γιατί οι μεγάλοι ούτως ή άλλως τα καταφέρνουν. Αλλά οι μικροί πρέπει να υποφεληθούν. Ποια θα είναι η στρατηγική σας γι' αυτό. Και τρίτο, ως παράδειγμα, στην Βαλτική, στο Φρίσα Χαφ, έχετε ένα εξαιρετικό κόλπο εκεί που υπάρχει. Και μπορεί κανείς και σε σχέση και με το Καλίνιγκραντ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά για την ε, διάβαση στο Μπιαλίστοκ πρέπει να δει κανεί ε, και την δυνατότητα αυτή και για την Πολωνία και για το Καλίνιγκραντ. Είναι σημαντικό να διαπραγματευτούμε με τους Ρώσους ώστε ο κόλπος του Φρίσα Χάφε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ αυτής της περιοχής και της Λιθουανίας και ιδιαίτερα για τις εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Φυσικά και εγώ θα της ευχηθώ κάθε επιτυχία. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μία πρόκληση, η Προεδρία σας ουσιαστικά έχει μία πρόκληση. Έχουμε αυτή τη νομική βάση, έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές και πιστεύω και εγώ ότι σε αυτό το φόρουμ της Καρακοβίας που είπατε θα πρέπει να δοθεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ο τομέας, ο κλάδος πρέπει να αποθεληθεί αυτής της νέας νομικής βάσης για να δημιουργηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετά το 2014, για την περίοδο 2014-2020. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εσωτερικό τουρισμό, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία Καλυψό που φίξατε και εσείς, που φέτος εκπνέει και είχε θετικές συνέπειες, πρώτα απ' όλα ότι κινητοποίησε έναν κοινωνικό τουρισμό. Και είδαμε και τις πτυχές της εποχιακής εργασίας. Στην Ευρώπη σήμερα, παρά τα όσα λέει ο Φιντάντσα, νομίζω ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε και τις ε, αγορές, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, Ευρωπαίων που ακολουθούν πολύ σημαντικές τουριστικές διαδρομές και θα πρέπει να προτείνουμε νέα θέματα, τα πολιτισμικά, την υγεία και άλλα. Θα πρέπει βέβαια να ενισχύσουμε ε, και το τομέα των ολοκληρωμένων ε, φυσικών πάρκων και ξέρουμε ότι Υπάρχει και η εργασία με τις νέες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει ε, ολοκλήρωση ε, των συστημάτων για μια πλήρη διαδρομή και αυτό πραγματικά απογοητεύει πολλούς. Καλό θα ήταν λοιπόν όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Το ίδιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα που έχουν. Κάθε φορά αντιμετωπίζουμε όταν πρέπει να εφαρμοστούν τα δικαιώματα, ε, την μεγάλη άγνοια του προσωπικού και την έλλειψη ενημέρωσης των επιβατών. Όλες επίσης οι πτυχές της αναρμόνισης της ποιότητας του εσωτερικού τουρισμού, της προσφοράς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα αυτά νομίζω ότι απαιτούν ε, εκπαίδευση και πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Ό,τι αφορά τον εξωτερικό τουρισμό θα σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να δούμε τις πλήρεις διαδρομές. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρώπη εργάζεται με κάποιους προορισμούς, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία. Ε, είναι πολύ εντοπισμένοι και περιορισμένες αυτές οι διαδρομές αντί να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση πιο πλήρων διαδρομών. Να μπαίνει κάποιο στη Γαλλία, να μπαίνει στο Παρίσι και να φτάνει στο άλλο άκρο της Ευρώπης για να δείξουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να προσφέρουμε πολιτισμική, γαστριμαργική κληρονομιά, αλλά και τη βιομηχανική κληρονομιά, όπως με επιτυχία πρότεινε ο πρόεδρός μας. Και να σας θυμίσω και εγώ το πρόβλημα ε, με τις βίζες, με τις θεωρήσεις διαβατήριο, όπου πάμε ακριβώς αυτό το θέμα μας θέτουν. Ε, είναι βέβαια ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο στη δική σας αρμοδιότητα, είναι υπερβαίνει το απαιδεία της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια ε, πολύ σημαντική χρονική περίοδο, ένα σημείο κλειδί για τον τουρισμό και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των τουριστών. Να μην πρέπει να στείνονται στις ουρές, ε, στις πρεσβείες ε, για να πάρουν ε, τη θεώρηση. Να υπάρχει ένα κομβικό σημείο που θα επιτρέπει την είσοδο αυτών των τουριστών και να μπορούν οι πρεσβείες να καταληφθούν αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά κυρία Υπουργέ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην εισήγησή σας. Δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω αν επιτρέπετε και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά στην αίθουσα ότι η ανάπτυξη του τουρισμού από πολλούς ε, δείκτες εξαρτάται από το επίπεδο ευημερίας των πολιτών, από τους στόχους και τις αξίες των ανθρώπων, επίσης εξαρτάται από την πολιτική κατάσταση στις διαφορετικές μας χώρες. Και όταν υπάρχουν πολιτικές ταραχές, τότε αποφεύγουν χώρες και περιοχές οι τουρίστες. Εξαρτάται όμως και από αποφάσεις ζωής ή μοιρές αποφάσεις. Όταν υπάρχουν θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα γεγονότα. Θέλω να αναφερθώ σε δείκτες που μπορούμε να επηρεάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά μια παράκληση τώρα μετά από αυτά κυρία Υπουργέ. Όταν πρόκειται για την ανάπτυξη του τουρισμού, τότε πρέπει σε πανενοσιακό ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια συμφωνία ενέκρινε για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας και Κορέας και Κορέας. Τώρα πρόκειται για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Όταν διαπραγματευόμαστε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες κάνουμε διαμακρόν λόγο πώς έχει η αγορά εργασίας, ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν για την αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Θα ήθελα να υποβάλω την εξής πρόταση όμως. Όταν ε, συζητούμε συμβάσεις και συμφωνίες με τέτοιες τρίτες χώρες και διαπραγματευόμαστε τέτοια πράγματα, πρέπει να απαντούμε το ερώτημα ποια επίπτωση έχουν όλα αυτά στην εξέλιξη του τουρισμού, στον ίδιο τον τουρισμό. Πώς επηρεάζουν τον τουρισμό όλα αυτά. Αυτή είναι η ερώτησή μου, αυτή είναι η παρεμβασή μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο τουριστικός τομέας σε σχέση με την οικονομία πώς θα επηρεαστεί. Θέλω να υποστηρίξω τους συναδέλφους εκείνους που προηγούμενα τοποθετήθηκαν και έκαναν λόγο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε σχέση με θεωρήσεις διαβατηρίων. Η Πολωνία είναι ένα καλό παράδειγμα κυρία Υπουργέ. Δεν αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα εξειδικευμένα, αλλά οι κανονισμοί διατάξεις του Σέγγεν είχαν μεγάλη τεράστια επίπτωση και για τον τουρισμό στην Πολωνία και θα έχουν και επηρεάζουν και τα πράγματα και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τουρισμός λοιπόν θα πρέπει να ανήκει στις αρμοδιότητες ε, του Επιτρόπου για τα εξωτερικά πολιτικά θέματα, διότι το Σέγγεν δεν είναι μόνο για τα θέματα ασφάλειας στην ίδια την Ευρώπη, αλλά και για την θετική επιρροή της προώθησης του τουρισμού. Ευχαριστώ. Uh, uh, Τέλος εγώ κύριε Πρόεδρε, ένα, δύο, κυρία Υπουργέ, συγγνώμη, ένα-δύο πράγματα. Θέλω να επισημάνω και εγώ ε, για τα όσα είπαν και οι υπόλοιποι για την οδηγία για ε, τα all inclusive πακέτα είναι ιδιαίτερο θέμα, διότι εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχουμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο. Μίλησε και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς ε, που γνωρίζει ότι είναι κομβικός ο ρόλος μας. Βεβαίως πριν κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να υπάρξει πρόταση. Ίσως θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ε, μία πλήρη αναθεώρηση της οδηγίας για τις all-inclusive ε, ε κρατήσεις, διότι όλα η οδηγία έχει προκύψει πριν να έχουμε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και πριν έχουμε πολλά άλλα πράγματα και επομένω ε, καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία αυτή είναι παροχημένη και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά τι θεωρήσει διαβατηρίων. Εγώ πάντα λέω αυτή την ιστορία που φτάνει κάποιο στο αεροδρόμιο του Χήθρου στο Λονδίνο ω ξένος τουρίστα που θέλει να επισκεφθεί τα θαύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και σας συναντά μία τεράστια πινακίδα που λέει «Καλώς ορίσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο» και η πρώτη ερώτηση του συνοριοφύλακα είναι «Πόσο σκοπεύετε να μείνετε». Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η αντιμετώπιση. Δεν ξέρω τι κάνει αυτούς τους ε, υπαλλήλους στα τελωνία και έχουν την ίδια ξυνήλα, αλλά φαίνεται ότι κανένας δεν τους ε, καλωσορίζει τους τουρίστες, ούτε τους κάνει να νιώσουν ευπρόσδεκτοι. Η αγγλική φιλοξενία. Το επόμενο θέμα το οποίο ήθελα να αναφέρω, ως τελευταία παρατήρηση, είναι αυτή η διάσκεψη στην Κρακοβία, την οποία αναφέρατε και είπατε ότι θα επικεντρωθεί σε θέματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι έχουμε να προσφέρουμε εμείς ε, ως Ευρώπη πριν να αρχίσουμε να μιλάμε για την ανταγωνιστικότητά μας ως Ευρώπη. Δεν πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ε, πλασάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κατάλληλο ε, τουρισμό όσο θα έπρεπε, διότι τα κράτη-μέλη με ζήλο διατηρούν τα δικαιώματά τους ε, στον τουρισμό στο παρελθόν. Ε, κατά την άποψή μου, πέρα από ορεινού όγκου και παραλίε, η Ευρώπη έχει πολύ περισσότερο να δώσει. Ο Μάικολ αναφέρθηκε στον ποδηλατικό τουρισμό. Εμεί έχουμε και βιομηχανική κληρονομιά, ευρωπαϊκή βιομηχανική κληρονομιά. Και εδώ ε, δίνονται δυνατότητε να αναπτύξουμε τουριστική βιομηχανία σε τομεί που ε, συνήθω δεν έχουν τουρίστε. Διότι βρίσκονται σε βιομηχανικέ περιοχέ, για παράδειγμα δεν νομίζω ότι πραγματικά μπορέσαμε να δράξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαιρία να πείσουμε τους τουρίστες να έρθουν να επισκεφθούν και να δουν αυτή τη μορφή της ιστορίας μας, αυτή τη μορφή του πολιτισμού που ανέφερε και η κυρία Γιάλα Σέντερ. Πρόκειται για ένα αμάλγαμα πραγμάτων που μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω στα οποία μπορούμε να δομήσουμε τον τουρισμό μου και νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Ταγιάννη ε, επιτέλους αρχίζει να αναγνωρίζει ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός είναι κάτι παραπάνω από τις Άλπεις και τις παραλίες και νομίζω ότι αυτό είναι ε, ζωτική σημασία ε, θέμα και θα πρέπει να το αναφέρουμε. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε. Σε ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ θερμά για όλες τις ερωτήσεις που διατυπώσατε. Διότι κάποια θέματα επαναλαμβάνονται βέβαια και ο χρόνος είναι περιορισμένος, είναι πεπερασμένος, γι' αυτό θα προσπαθήσω από κοινού κατηγοριοποιώντας, ομαδοποιώντας τις ερωτήσεις σας να απαντήσω στα θέματα. Πολλά ερωτήματα αναφερόντουσαν κυρίως στα θέματα και πτυχές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων όσον αφορά συνολικά τον τουρισμό και θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων. Εδώ θα ήθελα με κάθε πλήρη ευθύνη και υπευθυνότητα να πω ότι η Πολωνική Προεδρία την χρηματοδότηση και τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων τα θεωρεί τεράστια σημασία. Ιδιαίτερα αφορά το, η Πολωνία σε σχέση με την εισαγωγή του νέου συστήματος θεωρήσεων διαβατηρίων άσκησε μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας και γι' αυτό γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα εξιδίας πύρας, ώστε πραγματικά να προαχθεί η Ευρώπη και να μπορέσει να προωθηθεί ως δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες σε παγκόσμια κλίμακα. Και πέρα από αυτό θα συνεχίσουμε το έργο, τις εργασίες που αφορούν και έχουν ήδη ξεκινήσει και αναπτύχθηκαν και έχουν ως στόχο, αν είναι βέβαια πάντα δυνατόν, να μπορέσουν να τονώσουν και να προωθήσουν ώστε να υπάρξουν κοινέ διαδικασίες για τις θεωρήσεις διαβατηρίων για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή από ε, έξω ευρωπαϊκές χώρες. Και για το, τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια 2014-2020. Τα προγράμματα και τα πλαίσια αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας, ώστε να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για τον τουρισμό υπό την ευρύτερη έννοια, στο δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο και να μπορέσουν να υλοποιηθούν προγράμματα και σχέδια και μέσα από το πλαίσιο του σημερινού μηχανισμού χρηματοδότησης. Μέσα από αυτές τις δυνατότητες πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έχουμε ως ε, δυνατότητες σήμερα στις σημερινές δημοσιονομικές προοπτικές και μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες όπως αναφέρθηκε αλλά υπάρχουν δυνατότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην περιφερειακή πολιτική και για την πολιτική για τη συνοχή και για την πολιτική για την ανάπτυξη του χώρου της υπαίθρου. Παντού σε αυτούς τους τομείς υπάρχουν δυνατότητες ώστε κονδύλια, χρήματα να μπορέσουν να διατεθούν για τον τουρισμό υπό την ευρύτερη έννοια και σίγουρα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας εμείς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε το νέο πολιετές πλαίσιο σχεδιασμού 2014-2020 να κατατιστεί, να σχεδιαστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μετά για την οδηγία 314, την πιο σημαντική για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στα κράτη-μέλη. Περί πρόκειται εδώ. Εδώ είμαστε υπέρ μιας διαδικασίας ανανέωσης της οδηγίας, πλήρους ανανέωσης. Γνωρίζουμε ότι έχουν καθυστερήσει οι εργασίες, όμως όλα στοχεύουν στο σωστό προσανατολισμό. Το δυνατόν νωρίτερα να έχουμε μια επικαιροποίηση, ένα εξυγχρονισμό στην αναθεώρηση αυτού του κειμένου. Τον τελευταίο καιρό, στο τελευταίο διάστημα με την έκρηξη του ηφαιστείου καταδείχθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, ότι Πολλές ανάγκες πρέπει να αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν. Το φόρουμ, το βήμα για τον τουρισμό, επόμενη ερώτηση παρέμβασης Ευρωβουλευτού. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην πρώτη και κύρια προτεραιότητα που απορρέει από τη νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τουρισμό σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και την ενδυνάμωσή της. Τι εννοούμε υπό αυτό το πλαίσιο. Θέλουμε συζητήσεις να μπορέσουν να διεξαχθούν, συζητήσεις με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτυχθούν γύρω από τον άξονα των νέων τεχνολογιών και της τεχνολογίας που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο τουρισμός καλύτερα και την βέλτιστη προσπελασιμότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Αλλά όπως είπατε και εσείς ο ίδιος Πρόεδρε, αύξηση, αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει για τα προϊόντα τα τουριστικά να είμαστε ανταγωνιστικοί και στην εκπόνηση τέτοιων τουριστικών προϊόντων να μπορέσουμε Ω ως ε, κληρονόμοι της βιομηχανίας και της, του, της βιομηχανικής κληρονομιάς ως κληροδοτήματος να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε κυρίως να τονώσουμε αυτή τη συνιστόσα και τον Σεπτέμβριο όταν θα έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα για τον τουρισμό να μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το πολιτικό πολιτισμικό κληροδότημα της βιομηχανικής εποχής είναι τεράστια σημασία για μας και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο από τα κράτη-μέλη μας. Και στη συνέχεια όσον αφορά τη συμφωνία, συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και διαπραγματεύεται τα θέματα αυτά με τρίτες χώρες. Είναι φυσικά σημαντικό σε αυτό το πεδίο ο τουρισμός να λαμβάνεται και αυτός υπόψη και να δούμε πώς επηρεάζει τον τουρισμό μια τέτοια συμφωνία με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα στις ε, υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και την Μολδαβία, τη Μολδόβα. Ε, πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα πράγματα υπαρκώς υπόψη. Επίσης υπήρξε και μια ερώτηση του κυρίου Κράμερ που διατυπώθηκε σε σχέση με τον ποδηλατικό τουρισμό, τους ποδηλάτες και τον τουρισμό και τα βιώματα, την πείρα που έχουμε στην Πολωνία σε σχέση με τον τουρισμό αυτόν. Πρέπει να πω ότι εδώ και δύο χρόνια είναι προτεραιότητα για μας τους ίδιους τους Πολωνούς. Γνωρίζουμε ότι είναι μακροπρόθεσμος αυτός ο ορίζοντας και οι διεργασίες όσον αφορά τις σημερινές ε, χρηματοοικονομικές προοπτικές. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα για την ε, επέκταση των ε, ποδηλατικών δικτύων στις ανατολικές περιοχές και περιφέρειες. Να υπάρξουν τέτοιοι διάδρομοι και να καλυφθούν τα κενά στις υποδομές. Όμως ε, με επιτυχή τρόπο δραστηριοποιούμαστε κύριε Ευρωβουλευτά όσον αφορά την ανάπτυξη ε, του Ευρωποδηλατικού διαδρόμου 13 που είναι σημαντικός όσον αφορά την Πολωνία και που από πολωνικής πλευράς ε, θα ε, ε, υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική για την επισήμανση, σηματοδότηση αυτής της οδού και χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας με τις σημερινές ε, χρηματοοικονομικές προοπτικές. Είμαστε υπέρ του, της φραγίδας ή του σήματος ποιότητας. Πρέπει αυτό το πιστοποιητικό, η σήμα ποιότητας να ανταποκρίνεται φυσικά σε ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσει. Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις ή γραφειοκρατική επιβάρυνση που να συνοδεύει ένα τέτοιο σήμα. Θα πρέπει μία ένα ή δύο διαφορετικά σήματα να μπορούν να υπαρκέσουν για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και να υπαρκέσουν και να είναι αποτελεσματικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός και για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών μονοπατιών που δεν θα αφορούν μόνο μια χώρα αλλά αρκετές χώρες ευρωπαϊκά μονοπάτια όπως ανέφερε η κυρία Γιάλα Σέντερ είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα και αυτό να ληφθεί υπόψη. Έχουμε συγκεκριμένη πύρα που έχουμε συλλέξει σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης που υποστηρίχθηκαν και στηρίχθηκαν ιδιαίτερα όσον αφορά και τρίτες χώρες ε, το, της ΙΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία. Με μεγάλη επιτυχία συνδέθηκαν τέτοιες πρωτοβουλίες και πρέπει να συνεχιστούν πιστεύω. Κυρίως επειδή αυτές οι δραστηριότητες ε, αρθρώνονται μέσα στο πλαίσιο των μέτρων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται από πλευρά τη νέα ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι τα σημαντικότερα, τα ουσιοδέστερα σημεία τα κάλυψα με τι απαντήσει μου. Υπήρξε και μία άλλη παρέμβαση του κυρίου Κράμερ για τι. Ε, πλωτές ε, ποτάμιες μεταφορές. Αναφερθήκατε στο Frisches Χαφ επίσης της Βαλτικής. Ε, τυπικά και επίσημα οι διαπραγματεύσεις με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία ολοκληρώθηκαν και ελπίζω ότι οι πλωτές μεταφορές μέσω του Frisches Χαφ θα μπορέσουν να προαχθούν. Δεν θέλω όμως να αποκρύψω ότι εξακολουθούν και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και δυσκολίες όσον αφορά τη διαδικασία θεωρήσεων διαβατηρίων. Και αυτό συνολικά τις ε, πλωτές μεταφορές τις έχει επιβαρύνει. Ελπίζουμε ότι το δυνατόν γοργότερα θα υπάρξει μια συμφωνία επ' αυτών. Το πρόγραμμα Καλυψό για την Πολωνία ανήκει και αυτό μέσα στο πλαίσιο μιας σημαντικής προτεραιότητας σε σχέση και με την Ισπανία και Πορτογαλία για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα το οποίο την εποχικότητα την αντιμετωπίζει, προσπαθεί να την αντιμετωπίσει στον τομέα του τουρισμού αλλά αφορά και την διεύρυνση και επέκταση και άλλων μορφών κοινωνικού τουρισμού και γι' αυτό πρέπει να είναι εφικτό σε όλους τους ανθρώπους και πολίτες να, να ξεκουράζονται, να μπορούν να αναπαυθούν, να έχουμε και για τους ηλικιωμένους, για τα άτομα με μειονεξίες, για τους νέους δυνατότητες και για εκείνους που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες τουρισμού, ψυχαγωγίας, ανάψυξης, να μπορούν, αναψυχής με συγχωρείτε, να μπορούν να παρακολουθήσουν τέτοιες δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για τις παρατηρήσεις και ελπίζω ότι απάντησα σε όλα όσα αναφέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας στον τομέα του τουρισμού. Κάθε επιτυχία λοιπόν στην Πολωνική Προεδρία και ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα το επόμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση σας και που απαντήσατε τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Okay, can I... Λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσον υπάρχουν διάφορα, πρώτα απ' όλα. Αλλιώς να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρία μας θα λάβει χώρα εδώ στις Βρυξέλλες την 3η 30 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Και με αυτά και με αυτά σας εύχομαι καλές διακοπές. Ευχαριστή. Και εύχεται και στους διερμηνείς ο Πρόεδρος. Θέλω να ευχηθώ και στο προσωπικό. Καλές διακοπές. Ελπίζω να έρθετε όλοι ανανεωμένοι στα τέλη Αυγούστου. Ε, πέρα στις